Good afternoon, colleagues, and... Uh, Καλό σα απόγευμα και σα καλώ ορίζω στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ανάπτυξη αλλά και τη Επιτροπή Περιβάλλοντο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ καλ... για την ευκαιρία που έχουμε για μια τόσο σημαντική συζήτηση για του στόχου τη αναπτυξιακή πολιτική. Δύο λεφτά πρωτού ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να ζητήσω από του συναδέλφου μου τη Επιτροπή ε, Ανάπτυξη να αλλάξουμε την μέση ιδέα και να αναβάλουμε το θέμα το οποίο εκκρεμούσε την έκθεση Μπόλ να πάει τον Ιούλιο. Κάνουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή και μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε στην κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και τα υπόλοιπα σημεία της Επιτροπής Ανάπτυξης θα τα εξετάσουμε αύριο το πρωί στις 10.30. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, Καλώς ήλθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που εξ ονόματος Επιτροπής Ανάπτυξης μπορώ μαζί με τον κύριο Γιάβορ, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, να προεδρεύσω αυτή της ε, συνάντησης και μαζί με τους επικεφαλείς των τριών πάνελ για την ακρόασή μας που θα μας ε, θα διευθύνει τη συζήτηση για μερικά θέματα που είναι ιδιαίτερα νευραλγικά. Όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο στα Ενωμένα Έθνη θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικά, αποτελε, αποτελεσματικές κινήσεις για τον τομέα της εξάλληψης της ένδυας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι ένα πάρα πολύ λοιπόν, σημαντικό θέμα που μπορεί να προωθηθεί στα Ενωμένα Έθνη και τον επόμενο μήνα στην Αντισάμπαβα η Επιτροπή μας προετοιμάζει ένα φόρουμ για την ανάπτυξη που θα είναι και αυτό προετοιμασία για τη συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Και επίση εκπονούμε μια γραμμοδότηση τη επιτροπή Περιβάλλοντος για, το, για την COP21 στο Παρίσι, τη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τους επόμενους έξι μήνες, αν δούμε όλα όλες αυτές τις συνδιασκέψεις στην Αντισαμπέμπα, στην Νέα Υόρκη, στο Παρίσι είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα διεθνή εταιρική σχέση για ένα θεματολόγιο επέκεινα του 2015. Θα πρέπει να συνεργαστούν λοιπόν οι επιτροπές μας. Ξέρω ότι και η Επιτροπή εργάζεται για τα θέματα αυτά και ο κύριος Καρμένου Βέλα είναι παρόν μαζί μας σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ και η κυρία Μογκερίνη προσπαθεί <clears throat> να συντονίσει το έργο της Κομισιόν για όλες αυτές τις συνδιασκέψεις. Έχουμε λοιπόν το εκλεκτό αυτό πάνελ ομιλητών και προσβλέπω και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιαβόρ, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κύριε, Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής περιβάλλοντος, ασφάλειας και δημόσιας υγείας με μεγάλη χαρά. Σας προσκαλώ σε αυτή την κοινή ακρόαση για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως ξέρουμε, η έννοια της βιώσιμης ε, ανάπτυξης και των στόχων ε, της βιώσιμης ανάπτυξης γεννήθηκαν στην διάσκεψη του Ηνωμένων Εθνών το 2012 Ρίο Συνήκωση ως συνέχεια ε, των στόχων, των αντιξιακών στόχων της χιλιετίας για να απεικονίσουν τις προτεραιότητες για την ε, ανάπτυξη και να δημιουργηθούν ε, καθολικά εφαρμοστέοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και με αυτόν τον τρόπο σταματούν οι παλιές πρακτικές όπου είχαμε δύο Χωριστέ συζητήσει. Μία συζήτηση για την ανάπτυξη και μία χωριστή για τη βιωσιμότητα. Πιστεύω ότι με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ο ΙΕ ξεκαθάρισε ότι τελείωσε αυτή η περίοδος. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα χωρίς ανάπτυξη και αντίστροφα. Έχουμε μία και μόνη συζήτηση τους στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και πρέπει να βρούμε λύσεις και για τις δύο πλευρές του νομίσματος. Αυτή η ακρόαση είναι πολύ επίκαιρη. Το 2015 είναι κρίσιμη χρονιά για την βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της στόχιας με διάφορες παράλληλες διαδικασίες που ενισχύουν η μία την άλλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΙΕ. Η συμφωνία για την ε, παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2015 και πραγματεύσεις υπό τον ΟΗΕ για την σύμβαση για την ε, κλιματική αλλαγή, ε, το COP20, η διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 και η μακροπρόθεσμη πολιτική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά και πιστεύω ότι η η ατραπός που πρέπει να ακολουθήσουμε καθορίζεται από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι μια επίκαιρη και σημαντική συζήτηση αυτή που θα διεξάγουμε σήμερα και μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις του 2015 είναι το πώς οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα γίνουν τελικά αποδεκτοί σε επίπεδο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν το συνόλο της ε, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για να διαμορφώσει αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ευχάριστη και επικοδομητική συζήτηση σήμερα και ελπίζω αυτή η διάσκεψη να συνεισφέρει στην ε, εκκίνηση μιας νέας φάσης, μιας νέας περίοδου για την ανάπτυξη, πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα είδατε στην ημερήσια διάταξη ότι αυτή η δημόσια ε, ακρόαση έχει τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ε, παγκόσμια ανάπτυξη, την παγκόσμια στην ατζέντα για την παγκόσμια ανάπτυξη μέχρι το 2015. Ο Νταβόρ Στία ήταν εισηγητή του Κοινοβουλίου για το θέμα της ανάπτυξης με το 2015 ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Λίντα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά σε αυτό το πρώτο πάνελ της ακρόασης, όλους τους ομιλητές. Ε, έχουμε έξοχους ομιλητές, τον Επίτροπο για ε, Καρμένου Βαέλα, περιβάλλοντος την ειδική σύμβουλο του ΟΗΕ ε, Αμίνα Μοχάμεντ για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό το 2015 και τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ε, Θεματικού Συντονισμού και Πολιτικής Κλάους Ρουτχάουσερ από τη Γενική διάθεση ΤΕΒΚΟ. Θέλουμε να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι 4 και 45. Κάθε ομιλητής θα μας μιλήσει για 10 περίπου λεπτά και συνεχεία θα αφήσουμε κάποιο χρόνο για ερωτήσεις και μια συζήτηση. Ο ρόλος μου ως συντονιστή θα είναι να προσπαθήσω να κατευθύνω όλες τις ερωτήσεις, ε, να τις ομαδοποιήσω, ούτως ώστε να κάνουμε μια καλή συζήτηση και να μην ξεπεράσουμε βέβαια το χρόνο μας. Το θέμα το παρουσίασε ο πρόεδρος από την Επιτροπή ΔΕΔΕ και ο αντιπρόεδρος από την Επιτροπή ΕΜΒΗ ουσιαστικά. Γι' αυτό εγώ θα θέσω κάποια ερωτήματα. Πού βρισκόμαστε στη διαδικασία των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο εσωτερικό, αλλά και ποιος είναι ο εξωτερικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ΟΗΕ, ε, με τους εταίρους μας στη διεθνή κοινότητα. Πώς ε, προετοιμαζόμαστε και τα συμπράσματα του Συμβουλίου, ας πούμε, τι επιπτώσεις είχαν, τι πρόπτικες υπάρχουν για τη διάσκεψη στην Αντισαμπέμπα τον Ιούλιο. Πώς θα το στην, ε, και τι επιπτώσεις θα έχει στις οκορυφής του Σεπτεμβρίου. Πολλές ερωτήσεις. Θα ακούσουμε κάποιες απαντήσεις από τους ανθρώπους που είναι βασικοί παίκτες. Καταρχάς ο Επίτροπος, ο Περιβάλλοντος, Καρμέν Βέλ, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Λίντα, Μπένεντικ, Νταβόρ, όλους σας που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σε αυτήν την κοινή ακρόαση από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για να συζητήσουμε τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Όπως έλεγε και ο Νταβόρ, είναι μια πρώτη πρωτοβουλία εδώ και αρκετούς μήνες. Φέτος, το 2015, η διεθνής κοινότητα έχει μια ιστορική σημασία σε ευκαιρία να αλλάξει τον κόσμο και να θέσει τους αναπτυξιακούς ε, στόχους, όπως είπε και ο Γενικό Γραμματέας ε, του ΟΗΕ, ως στο δρόμο για την αξιοπρέπεια. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τη βιώσιμη ανάπτυξη που προστατεύει και τους ανθρώπους αλλά και τον πλανήτη μας. Φέτος έχουμε τρεις διασκέψεις, όπως αναφέρθηκε ήδη, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην Αντισαβέβα, για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Νέα Υόρκη και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι. Τρία γεγονότα λοιπόν, αλλά μία ευκαιρία, μία και μόνο ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχει μπροστά το κόσμο σήμερα. Μία και μόνη ευκαιρία που θα δώσει μορφή στον κόσμο μας και θα δείξει πόσο ο κόσμο μας θα είναι αύριο. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσουμε. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο προς τους στόχους τους αναπτυξιακούς της χιλιετίας. Σήμερα μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί ένα νέο κορίτσι να πηγαίνει σχολείο κάπου που παλιά δεν υπήρχαν σχολεία, δεν μπορούσε να πάει σχολείο. Να φανταστούμε ότι το ίδιο κορίτσι θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρισμό ή σε καθαρό νερό και ότι η οικογένεια του κοριτσιού αυτού να μην υποφέρει πια από ένδια. Με δύο λόγια, αυτό είναι το κοινωνικό δικαίωμα στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, σε καθαρό νερό και το οικονομικό δικαίωμα που έχουμε να μην υποφέρουμε από φτώχεια. Είναι ένα παράδειγμα για τους τρεις αυτούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως δεν πρόκειται μόνο για τους τρεις αυτούς πυλώνες, πρόκειται και για την διασύνδεση μεταξύ τους. Αυτό το νερό κορίτσι μπορεί να πάει σχολείο, γιατί δεν χρειάζεται πια να περπατήσει 5 χιλιόμετρα για να πάει να φέρει καθαρό νερό. Μπορεί να πάει σχολείο γιατί η οικογένειά του δεν υποφέρει από φτώχεια πια και άρα μπορεί να το στείλει στο σχολείο. Άρα γι' αυτό μιλάμε για το δρόμο προς την αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Συνεπώς, τώρα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στους πυλώνες αυτούς και στην διασύνδεση μεταξύ τους. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με το θεματολόγιο για μετά το 2015 μιλάμε για μεγάλες αλλαγές. Δεν μιλάμε μόνο για τη μείωση της στόχιας ή για την ε, σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος. Το Σεπτέμβριο στη διάσκεψη οι ηγέτες θα κληθούν να είναι πιο φιλόδοξοι και να δεσμευτούν για την ε, απάλληψη της φτώχειας σε όλες τις, τις μορφές και να πετύχουν τη συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη και για τις σημερινές γενιές αλλά και για τις επόμενες και ακόμα περισσότερο για τις επόμενες. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια φιλοδοξία που αλλάζει τον κόσμο. Και συγχρόνως έρχεται και μια νέα ευθύνη που έχει να κάνει με την εφαρμογή όλων αυτών μέχρι το 2030. Ξέρω ότι πρόκειται για φιλοδοξία που έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συμμερίζεται. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξή σας. Το θέμα τώρα είναι πώς θα τα καταφέρουμε. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να φέρουμε αποτελέσματα. Μια από τις μεγάλες καινοτομίε για το θεματολόγιο μετά το 2015 είναι η οικουμενικότητα. Όλες οι χώρες θα κληθούν να δράσουν, διότι όλες είναι υπεύθυνε και στο εσωτερικό τους πρέπει να δράσουν και να συνεισφέρουν προκειμένου οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν διεθνώς. Αυτή η επιμερισμένη ευθύνη είναι κάτι πολύ βασικό και η νέα εταιρική σχέση βασίζεται στην κινητοποίηση όλων των παραγόντων και των φορέων σε όλα τα επίπεδα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε το συλλογικό μας όραμα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλε τι κυβερνήσει και από τι αναπτυγμένε και από τι αναπτυσσόμενε χώρε, όπω επίση και από τι αναδυόμενε οικονομίε. Σημαίνει συγχρόνω συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τη κοινωνία των πολιτών, με την ευρύτερη έννοια. Στην καρδιά ε, της ε, σωστής εφαρμογής βρίσκονται όλοι και πρέπει να έχουμε και το σωστό προπολογισμό και τα σωστά εργαλεία και τις σωστές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποσαφήνισε αυτό στο συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου. Προκειμένου να έχουμε δικαίωμα στην ανάπτυξη πρέπει να εφαρμοστούν σωστά οι στόχοι. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής και να συμπεριλάβουμε το όραμά μας για μετά το 2015 σε αυτό. Για να προχωρήσουμε πρέπει να περάσουμε σε πολιτικές με τη συμμετοχή όλων και μεγαλύτερη συνοχή σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται να κατονίσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η φτώχεια και η βιώσιμη ανάπτυξη δρούν. Δεν πρόκειται μόνο για τον οικονομικό παράγοντα ή τον κοινωνικό, η φτώχεια φτωχεια επηρεαζει και την υγεία και το περιβάλλον. Η κατανάλωση ορυκτών επίσης που επιδοτούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες σημαίνει δισεκατομμύρια ευρώ δαπάνες το 2010. Φανταστείτε με αυτά τα χρήματα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τη φτώχεια και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι επιδοτήσεις αυτές δεν πηγαίνουν απαραίτητα στους φτωχούς. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και προστασία τους επίσης. Αυτό είναι μια επένδυση, δεν είναι κόστος. Άρα καταλήγει σε αποταμίευση και μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των εσόδων. Αν επενδύσουμε σωστά στη διαχείριση των υδάτων, αυτό σημαίνει ότι έχουμε χαμηλού κόστους πόσιμο νερό. Και από αυτό μπορούν να υποφεληθούν όλοι και να έχουμε κέρδη και στην υγεία στη συνέχεια. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσει το εμπόριο λευκής αρκός. Και αυτό να το κάνει σε συνεργασία με τους εταίρους της. Ο αγώνας αυτός θα βοηθήσει γενικότερα ώστε και παράνομα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή δεν χρησιμοποιούνται για να στηριχτεί άλλο λαθρεμπόριο ή να εμφανιστεί παρετέρω διαφθορά. Άρα είναι κέρδος για όλους και για την σωστή διακυβέρνηση και για το περιβάλλον και για το κράτος δικαίου. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν γιατί είναι σημαντικό. Όταν συζητούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε τους στόχους μας, σκεφτόμαστε και οι οικονομικές πολιτικές αλλά και μη οικονομικές πολιτικές. Χρειάζονται και οι μεν και οι δε επιπλέον πρέπει να δουλέψουμε από κοινού, να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας για να κρατήσουμε ψηλά τις φιλοδοξίες μας. Η αντίστοιχη βέβαια μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει να έχουμε καλά αποτελέσματα και το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη και το Δεκέμβριο στο Παρίσι. Θέλουμε φιλόδοξα αποτελέσματα από, όλα, από όλες αυτές τις συναντήσεις γιατί αν κάτι δεν πάει καλά ε, σε ένα από αυτά τα τρία υπονομεύονται και τα υπόλοιπα. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπουργοί των χωρών μελών μέχρι τώρα έχουν πετύχει πολλά προκειμένου να αναπτύξουν μία ενιαία ευρωπαϊκή θέση για τους στόχους μετά το 2015 που αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, αλλά αναγνωρίζει επίσης ότι πρέπει να υπάρξει νέα ε, δέσμευση υπέρ της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναπτύσσουμε τις ε, θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνοχή προκειμένου να πετύχουμε τον τριπλό στόχο, την τριπλή νίκη στην οποία αναφέρθηκα και νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της και στην εφαρμογή των στόχων του χρηματολογίου για μετά το 2015 και μέσω της εξωτερικής της δράσης αλλά και μέσω των ε, πολιτικών της στο εσωτερικό. Ήδη κοιτάμε να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε τη συνοχή των πολιτικών μας ανάμεσα στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους και την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με απασχόληση για όλους. Όσον αφορά το πακέτο για την κυκλική οικονομία, συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα το οποίο έχει άμεση σύνδεση με τους στόχους μας για μετά το 2015. Δημόσιες διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα για όλα αυτά τα θέματα και θα ήθελα να σας ζητήσω να συμμετάσχετε κι εσείς, να ενημερώσετε τους συμπολίτες σας και να τους ζητήσετε να συμμετάσχουν κι αυτοί. Και έτσι φτάνω στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους που βρίσκονται και στην καρδιά του θεματολογίου μας για μετά το 2015 και είναι και η βάση πάνω στην οποία βασίζονται τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε. Είναι κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί συνολικά. Επιπλέον, από την εφαρμογή πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και να λογοδοτούμε κάθε φορά όσον αφορά τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Πρέπει να εντοπίσουμε μής όπου βρισκόμαστε πιο πίσω, να λογοδοτούμε κάθε φορά και να δίνουμε κίνητρα και όθηση για αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο αναθεώρησης που να περιλαμβάνει όλους τους στόχους συνολικά. σε εθνικό, σε περιφερειακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ευημερία, η συμμετοχή όλων είναι ζωτική σημασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα έχει να παίξει έναν ρόλο κλειδί προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως ε, λογοδοτεί. Υψηλού επίπεδου επίσης πολιτικά φόρα θα αποτελέσουν τον ακρογωνίο λίθο για το εγχείρημα αυτό. Υπάρχουν άλλα φορά τα οποία μετρούν την πρόοδο που γίνεται όσον αφορά διάφορα επιμέρους στοιχεία του θεματολογίου. Αλλά αυτό το φόρουμ υψηλού πολιτικού επίπεδου θα συμπεριλάβει την αξιολόγηση όλων αυτών των επιμέρους φόρουμ. Συνεπώς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το φόρουμ υψηλού επίπεδου θα έχει τις σωστές πληροφορίες προκειμένου να μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα και κάθε χρόνο οι υπουργοί, οι υπεύθυνοι για τις τρεις πτυχές των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων θα συναντιούνται κάθε χρόνο και επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων κάθε τέσσερα χρόνια. Μόνο έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε την δέσμευσή μας και το ρυθμό μας προκειμένου να πετύχουμε τους βιώσιμού αναπτυξιακούς στόχους μέχρι το 2020. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους προσβλέπω στη συνάντηση του υψηλού επίπεδου πολιτικού φόρουμ τέλη Ιουλίου. Τέλος. Ελπίζω και είμαι πεπισμένος ότι μπορώ να βασιστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας στηρίξει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Μόνο έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι ο δρόμος προς την αξιοπρέπεια θα είναι ένα ταξίδι που θα το κάνουμε χέρι-χέρι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Commission. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την πλήρη επισκόπηση των περιβαλλοντικών πτυχών αλλά και της ανάγκης για τον αγώνα κατά της ένδυας και για τις τρεις διαστάσεις που εξήρατε των, της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεχίσουμε λοιπόν προηγουμένως. Βλέπω ότι έχουμε μεγάλη προσέλευση και κάποιοι στέκονται αλλά είναι όρθιοι, αλλά έχουμε κάποιες θέσεις οι οποίες νομίζω τώρα ότι είναι μεν κρατημένος για τους βουλευτές, αλλά εφόσον είναι ελεύθερες αυτές οι θέσεις, μπορείτε ίσως να κάτσετε. Μπορούμε να αφήσουμε στην πρώτη σειρά κάποιες θέσεις ελεύθερες για τους βουλευτές, αλλά καθίστε στις υπόλοιπες αν θέλετε, ώστε να παρακολουθήσετε πιο άνετα τη συνεδρίαση. Συνεχίζουμε τώρα με την Αμίνα Μοχάμετ, την ε, ειδική σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα για, την, για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης μετά το 2020. Αμίνα εξπέξει ένα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία του συνθετικού εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που αποτελεί και τη βάση <clears throat> για τις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουμε. Έχει μια τεράστια εμπειρία για τα θέματα αυτά, για την εφαρμογή των στόχων της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και μας ενδιαφέρει πολύ αυτά που έχει να μας πεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Συμπρόεδρο, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι παρούσα εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φτάσω σε εδώ. Ξέρετε ότι γίνονται οι διαπραγματεύσεις ακόμα που εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε να τελειώσει, να μια, τελειώσει σύμφωνια μέχρι την Παρασκευή για τη χώρα μου και συνεχίζονται ακόμα αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρόσκληση. Είναι πάντα μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερη υποστήριξη για ένα ημιτελές ακόμα έργο έχουμε δαπανίσει το μεγαλύτερο μέρο των τελευταίων τριών ετών σε μια προσπάθεια η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τι προκλήσει αλλά και τι επιδιώξει όλων για να μπορέσει να υπάρξει ένα θεματολόγιο το οποίο θα επιτύχει τον προσδοκόμενο στόχο, δηλαδή να υπάρξει πραγματικά αναζωγόνηση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, πάρα πολλά χρόνια μας έχει απασχολήσει, αλλά τώρα πια έχει οριμάσει εκφράσω την ε, εκτίμησή μου για το έργο που έχει γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ήδη πριν από δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να έρθει το θέμα αυτό στο προσκήνιο και η ανάπτυξη αλλά και το περιβάλλον με ένα συνεκτικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη βάση για μια εταιρική σχέση που μας φέρει προς τα εμπρός. Και θέλω να σας συγχαρώ όλους για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Μάιο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο στο χώρο αυτό και να προωθήσουμε και τις διαπραγματεύσεις της Νέας Υόρκης. Όπως είπε ο κύριος Φέλλα, είναι μια ιστορική στιγμή. Είναι μια χρονιά που θα πρέπει να έχει πολλές δράσεις. Δεν θα ξανά έχουμε ποτέ την ευκαιρία να έχουμε όλες αυτές τις δράσεις παράλληλα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ένδια και να έχουμε περιεκτική ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας ώστε να υπάρξει ένα θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν τα μέσα εφαρμογής επί τη βάση της συνδιάσκεψης της Δόχα και του Μοντερέι. Στις πρόσφατες συνεδριάσεις αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ένδυας και όλα αυτά μας οδηγούν σε μια οικουμενική ατζέντα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο για την αναπτυξιακή βοήθεια και τις ειδικέ της διατάξεις αλλά συγχρόνως και να αντιμετωπίσουμε τους υπόλοιπου πόρους που μπορούν να κινητοποιηθούν για να λειτουργήσει αυτό το θεματολόγιο βασιστήκαμε στους στόχους ανάπτυξης της χιλιετίας, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι στόχοι, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για ολοκληρωμένους και πλήρεις στόχους. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τώρα χάρη σε αυτό το σύνολο στόχων. Οι στόχοι της χιλιετίας επίσης και οι επικρίσεις που διατυπώθηκαν για αυτού του στόχου κυρίω σε ό,τι αφορά την οικειοποίησή του από τα κρατημέλη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμε. Καταλάβουμε ότι πρέπει τα κρατημέλη να παίξουν σημαντικότερο ρόλο, αλλά και οι εμπλεκόμενοι από την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει όλοι αυτοί να εμπλακούν. Βλέπουμε ότι οι περισσότερε επιδιώξει που θέλουμε να προωθήσουμε βρίσκονται στο έγγραφό μα. Πώ τώρα μέσα σε μια διαπραγμάτευση με 193 κρατη να παραμείνουν αυτά τα στοιχεία είναι δύσκολο. Είδαμε το τελευταίο σχέδιο για τα σχέδια μετά το 2025. Κάποια πράγματα λοιπόν μπορούν να προσθεθούν στο έγγραφο αυτό, αλλά για να κρατήσουμε το έγγραφο ως έχει είναι ήδη ένα επίτευγμα. Πρέπει να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία που ήδη τώρα υπάρχει. Στις τελευταίες μέρες, ακούγοντας απόψε 193 χωρών και προσπαθώντας να συμφωνήσουμε για τον τρόπο εφαρμογής μιας ατζέντα που είναι ήδη πολύ φιλόδοξη, είναι κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο εγχείρημα γιατί υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στον μικρότερο κοινό παρονομαστή κατά κάποιο τρόπο και να υποβαθμιστούν όλα αυτά. Υπάρχουν όμως μεγάλες προσδοκίες για αυτή τη συνδιάσκεψη από τον κόσμο που δεν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Έχουμε λοιπόν σε τρει εβδομάδε μια συνδιάσκεψη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θεματολόγιο και τον ε, Σεπτέμβριο θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα της χρηματοδότησης αυτής της ατζέντα. Αλλά και η συνεδριά της Λίμας και του Παρισιού για την κλιματική, ανα... κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της και αυτές είναι σημαντικό τμήμα του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης. Η Κριστίνα Φιγκέρα και εγώ πολλές φορές μιλάμε για το γεγονός ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε την γενική αυτή προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται και η κλιματική αλλαγή, αλλά και η αντιμετώπιση της ένδυας. Είναι για πρώτη φορά <clears throat> τόσο πολύπλοκα και τόσο αλληλοσυνδεόμενα τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο μας. Προσπαθούμε να βρούμε ένα θεματολόγιο λοιπόν το οποίο θα ανταποκριθεί στι αιτήσει που έχουν διατυπωθεί αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Σήμερα τα καυτά θέματα στην Ευρώπη είναι τα θέματα τη μετανάστευση κυρίω και όσο εσεί αντιμετωπίζετε το θέμα τη μετανάστευση, η δική μα ατζέντα προσπαθεί να βρει πώ θα σταματήσει αυτή η μεγάλη μεταναστευτική ροή αντιμετωπίζοντα τι αιτίε τη, αντιμετωπίζοντα την υποχρεωτική μετανάστευση που γίνεται σε πολλέ χώρε τη. Αφρικής. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μονάχα με αρνητικό τρόπο τη μετανάστευση. Είναι σημαντικό επίσης και το θέμα της απασχόλησης και για τις νέες γενιές. Η ενεργεία των νέων σήμερα και πάλι είναι κάτι χωρίς προηγούμενο σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι θα μπορούν να ενσωματωθούν στον εργασιακό χώρο. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι το εξή ότι όταν βλέπουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον αυτής της ατζέντα, θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση όχι μόνο σε αυτά τα οποία ξέρουμε αλλά και σε αυτά τα οποία θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της παραμέλησης και της μη επαρκούς επένδυσης σε ορισμένες από αυτούς τους τομείς. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν πράγματα ήδη σε αυτή τη γενιά για να σταματήσουμε την ένδια, αλλά υπάρχουν και τα θέματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά στο θεματολόγιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει όσο όλο και μεγαλύτερη <clears throat> δέσμευση και συμμετοχή όλων. Χαίρομαι λοιπόν για τις δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις συνεδρίες των G7 για την εγκύκλιο του Πάπα ε, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να διατηρήσει και την ορμή προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορούμε να είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αξιοπρέπειας και θα μπορούμε να πούμε σε όλους ότι σιγά σιγά θα πρέπει να γίνει αυτή η απαραίτητη μετάβαση και τονίζω ότι είναι μια μετάβαση. Οι στόχοι της χιλιετίας δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως και θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε, στο σύνολο των θεμάτων και όχι μονάχα σε μεμονωμένα θέματα. Το τελευταίο κομμάτι του δρόμου έχει σημαντικέ προκλήσει, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση τη ανάπτυξη εξακολουθεί το πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους να έχουμε ένα έγγραφο που να είναι αποδεκτό από όλους και να περάσουμε στην Αντίσα Μπέμπα με ένα κοινό έγγραφο. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φορολογικά θέματα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχουμε πολλά στοιχεία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν τα φορολογικά συστήματα. Η οι υποδομές είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ στην Ιγυρία προσπάθησα να υλοποιήσω του στόχου τη χιλιετίας και ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισα είναι τα προβλήματα υποδομών. Όταν προσπαθήσαμε να κοστολογήσουμε του στόχου τη χιλιετίας ήταν τεράστιο το κόστος γιατί έπρεπε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη υποδομή. Μου είπαν όχι μην το υπολογίσετε αυτό στους στόχου τη χιλιετία, αλλά πώ μπορεί κανεί να τα πετύχει του στόχου χωρί ηλεκτρισμό, χωρί δρόμους, χωρί. Ε, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν οι επιχείρησει και ο κόσμο τη αγροτική παραγωγή. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να υπάρξει δημιουργία υποδομή όχι απλώ, με βαθμιαίο τρόπο, αλλά η απαραίτητη αυτή δημιουργία ε, υποδομών που θα αλλάξει τι οικονομίε μα. Ποια λοιπόν είναι η πλατφόρμα η οποία θα μπορέσει να συνενώσει όλου του πόρου που χρειαζόμαστε. Σε πολλέ περιπτώσει, δεν έχουμε μονάχα την πεπαλαιωμένη υποδομή, αλλά υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί από φυσικές καταστροφές και από πολέμους. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία όχι να αντιμετωπίσουμε μόνο τα θέματα της ένδυας, αλλά να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πρασίνισμα των πόλεων μας και το τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με τις υποδομές αυτές σε ό,τι αφορά την υδροδότηση, την παραχή ηλεκτρισμού, το ενεργειακό μείγμα που χρειάζεται για να περάσουμε από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες ενέργειες και το εμπόριο είναι ένα κομμάτι του θεματολογίου, όλο και πιο σημαντικό. Πώς όμως μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν πιο ίσες συνθήκες στον χώρο του εμπορίου, ώστε όλοι να καταλήξουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία θετικού αθροίσματος, win-win. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία και αυτή δεν έχει ε, περατωθεί και τουλάχιστον δεν είχε περατωθεί χθε που ήμουν ακόμα στη Νέα Υόρκη. Όλοι αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει γίνει. Πριν από δυόμιση χρόνια Κανεί δεν ήθελε να αναφερθεί στην προβληματική αυτή. Υπάρχουν ε, πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των λιγότερο αναπτυσσομένων χωρών και ελπίζω ότι θα μπορέσει εδώ να υπάρξει μια λύση. Επίσης, έχουμε πολλές συμφωνίες οι οποίες δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά είναι σημαντικές για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι υπόλογα τα, κράτη μας, οι, οι επιχειρήσεις και οι άλλοι εμπλεκόμενοι και στις συζητήσεις που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι γίνεται σε επίπεδο χώρας και να αυξήσουμε την ε, παροχή εκθέσεων και αναφορών, να έχουμε όλο και καλύτερη συλλογή αξιοπίστων στατιστικών, να έχουμε καλύτερη ικανότητα να καταμετρούμε και να έχουμε ενδείκτες οι οποίοι δεν θα αφήνουν κανένα απ' έξω. Οι περιφερικοί φορείς επίσης που έχουμε θα παίξουν ένα σημαντικότερο ρόλο για να μπορέσουμε να συνθέσουν όλα αυτά τα στοιχεία Πρωτού φτάσουμε στο παγκόσμιο, στο οικουμενικό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο είναι ακόμα να εξελίξει. Εξακολουθούν να υπάρχουν εντάσεις για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου και αυτό δείχνει ότι πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό πλήρους επισκόπηση και αναθεώρησης. Πρέπει όχι μόνο να είναι ολοκληρωμένος αυτός ο μηχανισμός, αλλά να είναι και αφοσιωμένος σε αυτό το στόχο, σε επίπεδο χρηματοδότησης να έχουμε μια ειδική αφοσιωμένη παροχή εκθέσεων. Όλα αυτά τα θέματα εξακολουθούν να είναι εν εξελίξη, αλλά υπάρχει δέσμευση ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην Αντίσα με ένα εγγραφό περατωμένο που θα έχει συμφωνηθεί. Το μηδενικό σχέδιο, το σχέδιο εκκίνηση για το επέκεινα το 2025 είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο διαπραγματεύσεων αυτή τη βδομάδα και εδώ το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν παράλληλα άλλες αυτές οι διαδικασίες και χρησιμοποιούμε όλη την εμπειρογνωσία που έχουμε από τα κράτη-μέλη και από την κοινωνία των πολιτών και τι επιχειρήσει για να προωθηθούν αυτές οι διαπραγματεύσει. Νομίζω ότι υπήρξε μεγάλη επαφή μεταξύ των διαπραγματευμένων για μεγαλύτερη ευελιξία στις συζητήσεις αυτές. Το κείμενο αυτό στην εισαγωγή και το προήμιό του όπου αναφέρονται οι στόχοι για το πλαίσιο λογοδοσίας προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή την φιλοδοξία των 17 στόχων. Ξέρουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο όλα αυτά να προσγειωθούν και σε επίπεδο κάθε χώρας και εγώ φυσικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ. Θα πάψω να είμαι τμήμα αυτής της διαδικασίας και στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να επανέλθω στη χώρα μου στην Ιγυρία. Η Ιγυρία περνάει τις δυσκολότερες εποχέ στη ζωή τη τα τελευταία 8-9 χρόνια, έχει μια νέα κυβέρνηση που θέλει να τονίσει τη διακυβέρνηση, τι υποδομέ και την ασφάλεια. Αυτά μπορεί να κάνει μόνο μέσα σε μια τετραετή θητεία. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η δημοκρατία μα περιορίζει σε βραχυπρόθεσμους οριζόντε και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο του θεσμού ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτού του μακροχρόνιου κύκλου. Για μένα όμως είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Όπως είπε ο κύριος Καρμένου Βέλα για το μικρό κορίτσι. Στη δεκαετία του 1960 ήμουν ένα μικρό κορίτσι στην Ιγυρία όταν είχαμε την... όπου έχουμε πρόσφατα αυτή την κρίση του Μποκο Χαράμ. Έχω περάσει μια διαδικασία παιδείας, έχω ένα πιστοποιητικό γέννηση, έχω ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχω λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να ζω, να εργάζομαι στα Ενωμένα Έθνη. Άρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με αυτά τα κορίτσια που έχουν απαχθεί τα αγόρια τα οποία δεν γεννιούνται τρομοκράτε αλλά γίνονται σιγά σιγά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αιτία για όλα αυτά είναι η όξυνση τη ένδυα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι, εκεί είναι άμυρη ευθυνών η κλιματική αλλαγή. Η λίμνη Τσάντ που παλιά έπαινε κανεί και πήγαινε σε ένα πλοίο και μπορούσε να κινηθεί σε μεγάλε αποστάσει, τώρα πια είναι απλώ μια χαβούζα, έχει αλλάξει το νερό. Όλα αυτά μα έχουν φέρει στην κατάσταση που είμαστε. Πρέπει λοιπόν να ξαναδημιουργήσουμε τι κοινότητε μα στην Ιγυρία, να φτιάξουμε τι υποδομέ, να βοηθήσουμε του νέου να έχουν ένα μέλλον. Όλα αυτά είναι κάποιε προκλήσει οι οποίε πρέπει να αντιμετωπιστούν με το θεματολόγιο βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό δεν είναι μονάχα μια τεχνοκρατική άσκηση. Σημαίνει ότι όπω πηγαίνουμε σε επίπεδο κάθε χώρα, η εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε σε αυτή την αίθουσα, στου θεσμού μα, θα πρέπει να βγει από τα στεγανά και να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τι διάφορε ομάδε και τα διάφορα στρώματα ανθρώπων όταν προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα το θεματολόγιο του 2025 και πέρα από εκείνη την εποχή. Είναι πολλοί οι στόχοι και οι πολιτικές των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύπλοκες πολιτικές. Χρειαζόμαστε όμως στόχους οι οποίοι θα συνενώσουν όλους. Θα πρέπει όλοι μας να δούμε αυτούς τους στόχους ως μια επένδυση με μια προτεραιότητα στις χώρες μας. Οι χώρες μας δεν θα διατυπώσουν μόνες τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης θα έχουν κάποια δικά του σχέδια και θα χρειάζεται αυτό το πλαίσιο να είναι ένας κατάλογος που μας εξηγεί μέχρι πού φτάνει η εταιρική μας σχέση για να μπορέσουν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι να γίνουν πραγματικότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και θα είναι εφικτό τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια επανάσταση στη συλλογή των δεδομένων. Χρειάζονται όμω θεσμοί οι οποίοι να λειτουργούν καλύτερα, εταιρικέ σχέσει που να ξεπερνάνε το εθνικό επίπεδο, ώστε να έχουμε μια πιο επίκαιρη και ανθεκτική ε, συνεργασία με την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται θα πρέπει να δίνουν και τη δυνατότητα να μπορούν οι πολιτικοί μας να κάνουν έγκαιρες και σωστέ επενδύσεις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία σε σχέση με αυτό το θεμετολόγιο. Εγώ μίλησα με άτομα που είναι ειδικοί στην επικοινωνία για να τονίσω πώ θα πρέπει να τονίσουμε αυτή την έννοια του βιώσιμου. Στα, στη γλώσσα μου στην Ιγυρία δεν υπάρχει καν η έννοια τη δημοσιομότητα, Να μπορεί αυτή η ατζέντα να είναι κατανοητή στου λαού τη Αφρική, τη Άπο Ανατολή, τη Λατινική Αμερική κτλ να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι σημαίνει αυτό και να το οικειοποιηθούν, να καταλάβουν ότι είναι σημαντικό αυτό. Ο μηχανισμός λογοδοσίας επίσης είναι κάτι που θα πρέπει να το αποφασίσουμε στη Νέα Υόρκη αλλά περαιτέρω θα πρέπει να λειτουργήσει και σε τοπικό επίπεδο. Πώ θα πληροφορήσουμε καλύτερα του τους κοινοβουλευτικού μα, την κοινωνία των πολιτών, τι επιχειρήσει, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι μα είναι κατανοητοί. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν όλοι. όταν μιλάμε για την ε, ελεκτική λειτουργία των κοινοβουλίων πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί, αυτές οι δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τη δράση της εκτελεστικής εξουσίας και την επιτεύξη αποτελεσμάτων με τους προϋπολογισμούς που έχουν. Και θα έρθω τώρα στις εφαρμογές. Είδαμε τι κάναμε μέχρι στιγμής ε, σε μια μεταβατική περίοδο όπου υπάρχουν και φιλοδοξίες και προσδοκίες, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εφαρμογής. Η εφαρμογή όπου έχουμε Είχαμε ήδη πολλέ επιτυχίε, αλλά υπάρχουν και προβλήματα και κενά. Χρειαζόμαστε κάποιε δεξιότητε, χρειαζόμαστε θεσμική πλαισίωση, μία αναζωογόνηση για να ανταποκριθούμε στην παγκόσμια αυτή ατζέντα. Και αυτό αφορά όλου μα. Είναι μια, περιφε... παγκόσμια ατζέντα, μια περιφερειακή και μια εθνική ατζέντα. Στην κοινότητά μου, ποιο είναι ο πιο ευάλωτο αυτήν την κοινότητα και αυτό θα είναι η κλειδία λίθο για να, φτα... να τσεκάρω πού βρισκόμαστε όλοι ούτε ώστε να μην αφήσουμε κανένα πίσω, κανένα εκτό. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στον ΟΗΕ και βλέπουμε ότι οι πιο νέοι, ε, τα παιδιά, ε, οι νησιωτικές περιοχές είναι οι πιο ε, ευάλωτοι και θα προσπαθήσουμε να τους συμπεριλάβουμε. Η καθολικότητα επίσης είναι σημαντικό στοιχείο στην πολιτική και αυτό το κάνει ο ΙΕ πρόσφατα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ε, το τελευταίο που θα πω, είναι ο ρόλος ε, των ε, βουλευτών. Έχετε το κατάλληλο περιβάλλον, πρέπει να κάνετε κάποιες νομοθετικές προσπάθειες, ούτως ώστε να υπάρχει νομοθεσία που χρειαζόμαστε. να υπάρχει μια νομοθεσία που θα εξασφαλίσει ότι ένα κοριτσάκι θα έχει πρόσβαση στο σχολείο. Να έχουμε τους νόμους, ούτως ώστε να υπάρχει η απαραίτητη φορολογική μεταρρύθμιση. Ή επίσης να υπάρχει η αίσθηση ότι μας ανήκουν αυτά τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο. Ε, και να υπάρχει κατάλληλη παρακολούθηση. Μίλησα για τις ευθύνε, ε, το να μην αφήσουμε κανένα πίσω. Ε, θα πρέπει να βρούμε και νέους εταίρους ε, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί οι stakeholders. Συνήθως συζητούμε σε θημερές επίπεδο. Από από τη μία έχουμε τις επιχειρήσεις, ε, από την άλλη έχουμε την κοινωνία των πολιτών. Όλοι μαζί πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχει ο φόβος της κακοφωνίας, αλλά πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ε, για να βρούμε λύσεις. Ε, υπάρχει φόβος ότι μπορεί να αποτύχουμε. Πώς θα αποδείξουμε στον κόσμο ότι θα τα καταφέρουμε. Εάν δεν έχουμε ελπίδα όμως, τελικά τι νόημα έχει όλη η διαδικασία, τι νόημα έχει η προσπάθεια. Υπάρχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπων που αξίζουν αυτή την προσπάθεια, άρα πρέπει να προσπαθήσουμε. Θα πρέπει οι οι βουλευτές, να δουν τι κάνουμε εδώ ε, και επίσης ε, να δούμε τι κάνουμε σε επίπεδο χωρών. Ε, επίσης οι βουλευτές θα πρέπει να ταξιδέψουν από περιοχή σε περιοχή. Η δουλειά που κάνουν οι βουλευτές για την ενίσχυση των αδυνάτων δημοκρατιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Να συνευρεθούν, να συζητήσουν, να προκαλέσουν στον άλλον σε περιοχές που χρειαζόμαστε προσπάθεια ενίσχυση τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου, δικαιοσύνη κτλ. Πιστεύω ότι σε αυτή τη τελευταία προσπάθεια να ενισχύσουμε τα όσα έχουμε κάνει για να υπάρξει αξιοπρέπεια, ελπίδα, σεβασμός ο ένας για τον άλλο και σεβασμός βεβαίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αμίνα, thank you very much. You did use a little bit more than 10 minutes, but I think... Ευχαριστούμε, Αμίνα. Ε, ε περισσότερο χρόνο το 10 λεπτά, αλλά όλοι άκουσαν μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα μας είπα και άκουσα τον κόπο που χρειάστηκες περισσότερο χρόνο. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ποιότητας ε, των θεσμών. Δεν περιορίστηκε να μιλήσεις με κάποιες γενικές έννοιες, αλλά μας έδωσες ε, πολύ πρακτικά παραδείγματα από τη χώρα σου και πώς οι θεσμοί παίζουν ρόλο. Πιστεύω και ο Κλάους Ρουτχάουσερ ε, θα ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση, θα μιλήσει από τη σκοπιά της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ. Θα δώσω το λόγο στον Κλάους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος μετά από δύο τέτοιους ομιλητές που ήταν τόσο πλήρης. Επίτροπε, αμίνα. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς, χαίρομαι που έχουμε και τις δύο επιτροπές εδώ για αυτό το θέμα παρούσες. Στο μέλλον, καλό θα ήταν να συμμετάσχουν περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γιατί αυτό για το οποίο συζητάμε είναι κάτι πολύ ευρύ. Και ξέρουμε ότι η συνοχή των πολιτικών είναι κάτι πολύ σημαντικό για να εφαρμόσουμε την ατζέντα για τους ε, στόχους αυτούς. Να μιλήσουμε δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πολιτικές και όλες οι πολιτικές να είναι ε, για να φτάσουμε σε αυτό που επιθυμούμε. Είμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου είναι στη Νέα Υόρκη με του συναδέλφου από τα κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι οι συζητήσει είναι δύσκολε, κυρίω ε, σε αυτή τη φάση. Είναι πολύ δύσκολο για το πώ θα εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Εκεί γίνονται οι διαπραγματεύσει. Όπω είπε η Αμήνα και άλλοι, η διάσκεψη οι διασκέψεις μάλλον, ε, είναι αλληλένδετες που θα γίνουν φέτος. Ε, και το να πετύχουν όλες είναι σημαντικό για να πάμε καλά στην Νέα Υόρκη. Το ίδιο ε, συμβαίνει και για τις επόμενες δύο διασκέψεις. Η επιτυχία στην μπέμπα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή. Οι συνάδελφοι στη Νέα Υόρκη δουλεύουν νυχθημερών για να πετύχουν συμφωνία, αλλά όπως είπε και η Αμήνα σήμερα το πρωί αλλού, το γεγονός ότι οι συζητήσεις είναι δύσκολες σημαίνουν ότι όλοι τις παίρνουν πολύ στα σοβαρά και ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον παγκόσμια. Αυτό είναι καλό σημάδι. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κλείσει τη συμφωνία αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ακόμα μια αποτυχία. Είναι σημάδι ότι πραγματικά όλοι δεσμεύονται να πετύχουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και η Κομισιόν, αλλά και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη είναι πολύ θεσμευμένα. Αν διαβάσετε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το Μάιο ή αν διαβάσετε το, το ψήφισμα ή τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλέ θεσμεύσει, αλλά αν συγκρίνετε αυτά που είχαμε στι πρόσφατε κοινοποίησει τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου με αυτό που υπάρχει τώρα επιτάπητο στη Νέα Υόρκη, θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφορά, μια ποιοτική διαφορά. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και τους ε, πολιετής ε, στόχους, τους ε, στόχους συγγνώμη, της χιλιετίας, αλλά και τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, τους έχουμε πάλι παράλληλα, τους έχουμε συγχωνεύσει. Και αυτό το το κάναμε μετά από μεγάλη επιμονή. Το πετύχαμε, πετύχαμε αυτή τη συγχώνευση μετά από μεγάλη επιμονή. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη φάση τη εφαρμογή. Και θα επανέλθω σε αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήδη μπορούμε να φανταστούμε, να προλάβουμε, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε αμέσω να, τα να προλυαίνουμε το έδαφο. Εάν κοιτάξετε την ανακοίνωσή μα του 2014 και τη συγκρίνετε με το κατάλογο των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων, θα δείτε ότι υπάρχουν εντυπωσιακό είναι, αλλά υπάρχουν πολλές επικαλύψεις. Δηλαδή όχι μόνο έχουμε πλήρη ατζέντα από την αρχή, αλλά καταφέραμε ε, η ανοιχτή ομάδα εργασίας να τον αναγνωρίσει αυτό. Οι μεγάλες προκλήσεις όμως ε, είναι μπροστά μας και η πρώτη είναι η Αντισαμπέμπα. Γιατί θα πρέπει να αποδείξουμε ότι τα μέσα εφαρμογή που θα βρούμε ως κοινέ δεσμεύσει όλες εμείς οι χώρες από όλο τον κόσμο θα είναι αρκετά φιλόδοξα και επαρκή για να εφαρμοστούν οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι. Ε, Αλλιώ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε τα μέσα για να εφαρμόσουμε του βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου ε, στην Αντισαμπέμπα. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη. Καταφέραμε και να μην το υποτιμήσουμε ότι ε, επιβεβαιώσαμε τους στόχους 0.7 ε, και είμαστε η μόνη περιοχή του πλανήτη που πήρε αυτούς τους, ε, αυτές τις δεσμεύσεις. Μην το ξεχνάμε και δεν είμαστε μόνο αμυντικοί, γιατί εμείς κάνουμε, κάνουμε πάρα πολύ καλή προσφορά και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Και Υπάρχουν και άλλες ε, μεγαλύτερες ροές για την εφαρμογή που μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Επίσης, αυτό ήταν το πρώτο χρηματοδότηση. Δεύτερον, πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, η πόροι για να εφαρμόσουμε τους στόχους. Η Αμίνα ε, μίλησε για τον ιδιωτικό τομέα. Ε, ο ιδιωτικός τομέας κινητοποιείται μόνο αν υπάρχουν σωστές πολιτικές. Ε, τα λεφτά τότε θα βρεθούν. Μόνο τότε θα βρεθούν. Γιατί ενδιαφέρονται στο βαθμό που υπάρχουν σωστέ πολιτικέ. Με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και με τι δεσμεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην Αντισαμπέμπα φιλόδοξα και να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε καλή προσφορά και το G77 θα, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εμείς στην άμυνα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αλλάζουμε ε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Από την διάσταση βορράς-νότος ε, μιλάμε για μια παγκόσμια διάσταση. Μιλάμε για μια καθολική ατζέντα, για την καθολικότητα της, των στόχων της ατζέντα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το προσπίσουμε και να δούμε και τι επιπτώσεις έχει. Η καθολικότητα τι σημαίνει ότι στι αναπτυγμένε χώρε θα πρέπει εμεί επίση να εφαρμόσουμε αυτή την ατζέντα. Και όπω είπα στην αρχή, το θέμα δεν είναι η κοινότητα μόνο που ασχολείται με την ανάπτυξη και, και το περιβάλλον να εφαρμόσει αυτού του στόχου. Όλοι θα πρέπει να του εφαρμόσουν, όλο το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε με τον τρόπο που οι κυβερνήσεις μας αλλά και η κοινωνία των πολιτών κατανοούν την έννοια της καθολικότητας, οικουμενικότητας. Και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στον τρίτο κόσμο, θα πρέπει να δώσουμε εμείς το παράδειγμα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών και τους μη κρατικούς φορείς. Ε, για την κλιματική αλλαγή, για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μια και είπα ότι θα Είμαι σύντομο. Τελειώντα, να σα πω τι θα κάνουμε τι επόμενε εβδομάδε. Είναι να κρατήσουμε ψηλά ε, τη φιλοδοξία, αλλά και να είμαστε και ρεαλιστέ παράλληλα. Δεν έχει νόημα να είμαστε υπέρ των δέων ε, φιλόδοξοι. Θα πρέπει, να βρούμε, θα τη σωστή φιλοδοξία ανάμεσα στο ότι είναι ρεαλιστικά εφικτό και στο ότι μπορούμε να κάνουμε και εμεί οι ίδιοι. Χρειαζόμαστε επίση να υπάρχει ε, φιλοδοξία και τέτοιε διασκέψει. κράτη-μέλη, αλλά και στην ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών, του Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμά του διαπραγματευτέ να έχουμε αυτή την υποστήριξη. Να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να διατρανώσουμε αυτή τη φιλοδοξία, αν έχουμε αυτή την υποστήριξη πίσω μα. Thank you, Ευχαριστούμε, πολύ, Κλάους. Ήσουν πολύ ξεκάθαρος για το πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων με τις διαπραγματεύσεις και πώς θα μπορούσαμε ρεαλιστικά να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Συζήτηση τώρα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Βέλα και καταλαβαίνω ότι πρέπει να μας αφήσετε. Ε, πάντως η συνεισφορά σας σίγουρα ήταν πολύ σημαντική και τις ιδέες σας θα τις χρησιμοποιήσουμε και στη συζήτηση. Απευθύνομαι τώρα στους ευρωβουλευτές για ερωτήσεις. Έχω πέντε τουλάχιστον στον κατάλογο ομιλητών. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό καθένας, παρακαλώ, για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Ο Σάρλς Γκέρενς είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους στόχους, έτσι όπως μας τους παρουσιάσατε, με τόσο ενθουσιασμό, με τόση αποφασιστικότητα. Όμως, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν έχουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε για τη χρηματοδότηση. Τα χρήματα χρειάζονται, έλεγε ο Woody Allen, αν μη τι άλλο για οικονομικούς λόγους. Οπότε, οι αμφιβολίες μου έχουν να κάνουν με το εξή. Στο Μότρα είχαμε ήδη θέσει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τηρήθηκε όμως. Ανανεώθηκε το 2005 τον ε, γράψαμε, τον χτυπήσαμε στο μάρμαρο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης δεν ακούστηκε τίποτα το δεσμευτικό. Μιλάμε για το 2030 και μετά το στόχο δηλαδή του 0,7% χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, ξεκινάμε με τη φήμη εκείνων που ανακοινώνουν, που λένε, υπόσχονται, αλλά δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Και εδώ δεν τα βάζω τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο με τις χώρες μέλη, γιατί ορισμένες χώρες μέλη είναι παραδειγματικές, άλλες όμως είναι δράμα. Δεν καταφέρνουν τίποτα και με την κρίση ακόμα λιγότερο. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς όμως θα πρέπει να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη μία-μία να μας πούν γιατί δεν τηρούν τους στόχους τους και οι υπόλοιπε γιατί τους τηρούν τους στόχους τους, γιατί τα καταφέρνουν. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο είμαι πολύ σκεπτικιστής είναι ότι δεν βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα ποια χρήματα θα, χρηματο... Ε, γιατί ποια κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν το περιβάλλον, ποια θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Αυτά που θα πάνε στην ανάπτυξη, μήπως τελικά θα χρηματοδοτήσουν το κλίμα. Είχαμε, θα θυμόσαστε, με την κυρία Εντιγκάρτε, πολύ δυσάρεστη συζήτηση από αυτού και είναι κρίμα που ο Επίτροπος Βέλα μόλις έφυγε, αλλά θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ξεκάθαρα ποιος θα κάνει τι, σε ποιο τομέα. Τέλος. Και πάλι σε σχέση με τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών Ανάπτυξης. Έγινε κάτι μετά και αυτό ήταν η μείωση 43% ε, σε μία χώρα μέλος. Τα συμπεράσματα δηλαδή δεν στέκουν πια. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Και ο μόνος τρόπος για να βγούμε από τα διέξοδο είναι να επιμείνουμε για εναλλακτικά μέσα και ανοτόμα χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορεί να προστατεύσει ακόμα την τιμή της πηγαίνοντας στην Αντίσα Μπέμπα λέγοντας ξεκάθαρα τι θα κάνει. Όχι με λόγια, σε πράξεις. 100 εκατομμύρια πού θα τα βρείτε για το 2020. Πείτε το μου. Με κάθε σεβασμό που έχω για σας κύριε Ρόντι Σάουσερ λέτε ότι όταν καθοριστούν οι στόχοι θα βρεθούν τα χρήματα. Ελπίζω να έχετε δίκιο, ελπίζω. Αλλά από την εμπειρία που έχουμε εμείς μέχρι τώρα τόσο συχνά μας κορόιδεψαν που ειλικρινά είμαι πολύ επιφυλακτικός. Γι' αυτό σας λέω. Η Μαρία Χόιμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, ομιλίες σας, κυρία Μοχάμετ. Είπατε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια συνέχιση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Αλλά πώς θα καταμετρηθεί η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων και πώς θα υπάρξει η εποπτεία τους, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάτε για τα δεδομένα. Προφανώς θα συμβάλλουν, αλλά παραμένει και ένα σύνολο από ερωτήματα. Ό,τι θα επιτευχθεί λοιπόν στην Αντίσα Μπέμπα θα πρέπει να συναρμόσετε με του στόχου του 2025. Όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να υποπτεύεται από κοινού γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Μιλήσατε για την επικοινωνία, είπατε ότι μιλήσατε με άτομα που είναι ειδικοί στα θέματα επικοινωνία. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε συγκεκριμένε ιδέε για μια καλύτερη επικοινωνία με τον έξω κόσμο που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Και ένα τρίτο ερώτημα προ τον ε, Επίτροπο Βέλα κανονικά θέλω να το θέσω, αλλά δεν είναι, πολύ, δεν είναι παρόν. στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Και υπάρχει πολλές φορές η επίκριση ότι ο ιδιωτικός ε, τομέας αναλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των στόχων αυτών μετά το 2025. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι πράγματι οι επιχειρήσεις θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ένδυας και όχι μονάχα για μεγαλύτερη κερδοφορία. Πρέπει να υπάρξει η καλύτερη λογοδοσία για τα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, το καθαρό νερό θα πρέπει να είναι κάτι που το θεωρούμε ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι απλώς μια καλή και ζουμερή επιχείρηση για τους ε, εργοδότες και τις επιχείρησεις. Η Heidi Ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα πριν υπουργό της χώρας στην οποία αναφερθήκατε, πριν υπουργό ανάπτυξη που αναγκάστηκε κατά 43% να μειώσει την αναπτυξιακή της ε, βοήθεια και είμαι γι' αυτό απογοητευμένη τελευταίος υπουργός. Και η ερώτησή μου ακολουθεί αυτά που είπε και ο κύριος Γκέρενς. Και εκείνο είναι τέσσερις υπουργός ανάπτυξης που για το 1% του ΕΠ. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για την εφαρμογή και για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Δεν νομίζετε ότι είσαστε υπερβολικά απολογητικός, κύριε Ρούντι Σάουζερ, όσον αφορά τον ρόλο μας και τις δεσμεύσεις μας που δεν τις φέρουμε σε πέρας. Έχει αποδειχτεί και από τις στατιστικές που είχαμε τέλη Μαΐου από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Εξηγήστε μας λοιπόν σας παρακαλώ λίγο περισσότερο πώς θα μπορούσε να πιέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αν μη τι άλλο να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Και βέβαια και χρειαζόμαστε καινοτόμα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, αλλά αυτό επιπλέον από τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί. Συνεπώς και σε εσά κυρία Μίνα Μοχάμετ, η καινοτόμα χρηματοδότηση τι μορφή παίρνει στα πλαίσια της διάσκεψης του Αντίς Αβέμπα και πριν από την συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Έκα. Ευχαριστώ. Δυστυχώ πρέπει να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Γκέρνς. Εγώ νομίζω ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη πραγματικά μια βιώσιμη πολιτική Έχουμε πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πεινούν σε αυτόν τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως και στο παρελθόν, δίνουμε τεράστια ποσά που οδηγούν σε σπατάλη ουσιαστικά. Πάνω από 50% της παγκόσμιας παραγωγής ε, ε, δημητριακών πηγαίνει για τη διατροφή ζώων. Καταστρέφουμε τροπικά δάση για να μπορέσουμε να έχουμε ε, χώρο για την καλλιέργεια. Υπάρχει τεράστια κατανάλωση ζωικών πρωτεϊών στα αναπτυγμένα κράτη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει τεράστια πείνα και ένδια. Κάθε δύο δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ δεν βλέπω να υπάρξει καμία στάση υπέρ της ε, βιώσιμης ανάπτυξης από τον ιδιωτικό κόσμο της επιχειρήσης είναι απλώς ένα σύνθημα. Θα πρέπει να βρούμε καλύτερους διάβλους για να προωθηθεί αυτή η πολιτική ώστε να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τον τρόπο διατρο... για όφελος αυτών που διατηρούν την παραδοσιακή της διατροφή στις αναπτυγμένες χώρες. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομες, λέω πρόεδρε μου, σε ένα λεπτό. Κύριε Σράντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη. Okay. Θα πρέπει να είμαστε θετικοί. Να έχουμε μια θετική στάση, όπω είπε και ο Επίτροπο. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να είμαστε αρνητικοί, αλλά το βασικό ποιο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να πετύχουμε, πώ μπορούμε να είμαστε θετικοί. Γι' αυτό συναντιόμαστε εδώ. Γιατί μιλάμε για την ενέργεια, για του φυσικού πόρου, και υπάρχουν πολλές εταιρείες έτοιμες να επενδύσουν και να διαθέσουν πόρους. Μιλάμε για πολλά πράγματα που η Ευρώπη, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν αντιμετωπίζουμε ήδη. Επίσης θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία στην πολιτική και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα κονδύλια που έχουμε. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και να θέσω ε, ένα ερώτημα στην κυρία Μαχάμεντ. Ίσως ε, δεν ε, είναι εντό θέματος, αλλά μίλησατε για την Ιγυρία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την δίωξη των χριστιανών στην Ιγυρία. 450.000 οικογένειες χρειάστηκε να φύγουν επειδή ήταν χριστιανοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να το δούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε θετικοί. Το βασικό είναι πώς μπορούμε να βοηθούμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ, κύριο Φλόρεντ. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε χρόνο τα ίδια ακούμε και πάλι τα ίδια πράγματα καταλήγουν. Το θέμα είναι το θέμα της ε, εφαρμογής αυτών των μέτρων. Αυτά ακούμε κάθε φορά, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κατάσταση στον κόσμο είναι όπως έχει. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της, του Ισλαμικού κράτους και της Ουκρανίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια ώστε να έχουμε μια πραγματική κοινή πολιτική για την ανάπτυξη, μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση. Θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας στην πλάστικα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αναρωτιέμαι αν είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε αυτούς τους στόχους με σαφή τρόπο. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Θα πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτούς που είναι στις χώρες προέλευσής και μεταναστεύουνε. Εμείς στη Χάγη στο Βερολίνο μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε, αλλά θα πρέπει κύριε Πρόεδρε και με κόψτε, θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει στις χώρες αυτές. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι προτάσεις θέλουμε, αλλά πώς θα τις εφαρμόσουμε στις χώρες αυτές από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αυτό είναι το ερώτημα. Λίντα, you θέλεις και εσύ να θέσεις ένα ερώτημα. Ευχαριστώ. Για το ίδιο θέμα. Ότι είχαμε τι ημέρε τη Ευρωπαϊκή Ανάπτυξης, κάποιοι από τους βασικούς εταίρους μα μου είπαν ότι ανησυχούν για τους 160 στόχους. Όταν όμω ε, είδαν τους στόχους αυτούς κάποιοι, είπαν ε, τι θα υπογράψει ο Μάρτιν. Το θέμα είναι Πώς θα το, συζητήσουμε εμείς που ασχολούμαστε με το περιβάλλον ή με την ανάπτυξη και όχι οι υπόλοιποι. Και μία ερώτηση προς την αμήνα. Οι κυβε, κυβερνήσεις χρησιμοποιούνται μία checklist, είπατε. Το βασικό είναι ότι μπορεί να υπάρξει αποδυνάμωση των στόχων αν χρησιμοποιούν αυτά τα checklist οι κυβερνήσεις. Και εγώ μια ερώτηση το ίδιο μήκο κύματο. Ακούσαμε τον Επίτροπο Βέλλα που απαρίθμησε πολλά στοιχεία, πολύ σημαντικά. Μίλησε, α πούμε, για τη σημασία της προστασία των ζώων. Παγκόσμια. Που ίσως δεν εντάσσεται ή δεν απεικονίζεται καλά σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα έχουμε τόσα πολλά άλλα θέματα. Το ερώτημα είναι πώ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολυάριθμες προτεραιότητες. Στην σύνοψη που μας έκανες, μας είπες ότι είναι, καλό να έχουμε έξι πυλώνες, ας πούμε. Το ερώτημά μου είναι το εξή. σε αυτές τις δια, κυβερνητικές διαπραγματεύσεις, κατά πόσον θεωρούνται και οι έξι αυτοί πυλώνες ε, προτεραιότητες. Αμίνα, ε, θα ήθελα να πάρεις πρώτο τον λόγο και να απαντήσεις στις πολυάριθμες αυτές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί με τις ρωτήσεις αυτές μας ε, βοηθάτε να εστιάσουμε καλύτερα ε, στα όσα κάναμε. Στη Νέα Όρκη μερικές φορές ε, οι συζητήσεις γίνονται αποσυνδεδεμένα από αυτούς που θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Για την έκθεση follow-up σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Ξέρουμε από τους στόχους της ότι, ότι πόρα απέχουμε από το να μπορούμε να πούμε άνετα πετύχαμε αυτά. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά κενά στα δεδομένα από διάφορε χώρε και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, με του στόχου του 2016 θα πρέπει να ενισχύσουμε του θεσμού, σίγουρα. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Θα πρέπει να επενδύσουμε στου θεσμού, ώστε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Ε, το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου συζητάει το ποιο θα είναι το πλαίσιο για την έκθεση follow-up. Και θα πρέπει να ξεκινήσει τι εργασίε του κανονικά την επόμενη εβδομάδα. Ε, αλλά θα ολοκληρώσει του χρόνου και οι στατιστικές επιτροπές στην συνεχεία θα ετοιμάσουν δείκτες ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη έμφαση στο να εξασφαλίσουμε ότι και η χρηματοδότηση τη ανάπτυξη και η στόχοι μετά το 2015 συνάδουν μεταξύ του. Αν κοιτάξουμε τα μέσα εφαρμογή για, για το στόχο 17, θα δείτε ότι αντικατοπτρίζονται στο έγγραφο για τη χρηματοδότηση. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή αυτά που λέμε στη, στο ένα επίπεδο να αντικατοπτρίζονται στην άλλη. Σε ό,τι αφορά ανακοινώσει υπάρχουν πολλά πράγματα. Η κοινωνία των πολιτών έχει πάρα πολλά δίκτυα ε, και μας ε, και έχουν και καλές ιδέες για το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο για την ατζέντα αυτή. Θα προσπαθήσουμε εμείς να γνωστοποιήσουμε παντού αυτούς τους στόχου. Είναι πολύ σημαντικό ε, να το κάνουμε αυτό σε επίπεδο χωρών, ειδικά όταν να φτάσουμε στο επίπεδο της Ε, και ο ΙΕ εργάζεται επί του θέματος αυτού σε συνεργασία με κάποιες χώρες και με τους εταίρους μας. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα που αναφέρατε. Θέλουμε να έχει μεγαλύτερο ρόλο ο ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι ανησυχίε που υπάρχουν. Όπου πολλοί από την κοινωνία των πολιτών, πολλέ από τι κυβερνήσει του G77 ανησυχούν ε, για το πώ έγιναν ε, όλε οι προσπάθειε στο παρελθόν και σε ποιο ε, σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε τον κατάλληλο έλεγχο, ούτως ώστε να γίνουν σοβαρά οι προσπάθειες. Ε, ήμουνα την περασμένη εβδομάδα μια-δυο μέρες στον ΩΣΑ που έκαναν ε, μια τεράστια συνεδρίαση για την ευθύνη των επιχειρήσεων. Το αντιμετωπίσουμε τώρα από, το, τη σκοπιά του επιχειρηματικού μοντέλου. Ποιο είναι το μοντέλο αυτό, ούτως ώστε να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δείκτες ε, θα μας βοηθήσουν να μετρήσουμε αυτή την ε, προσπάθεια και θα πρέπει ε, να καθίσουν οι κυβερνήσεις στο τραπέζι κτλ. Και συνεχεία σε επίπεδο χώρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Ε, θα πρέπει και η κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις κτλ. να λογοδοτούν, ούτως ώστε όλοι αυτοί να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Ε, και στο μηχανισμό follow-up και στην δημιουργία των δικτών. από τα εκατομμύρια στα δισεκατομμύρια. Γίνεται μια δουλειά με αυτή την πρωτοβουλία. Ε, και υπάρχουν και άλλοι πόροι ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Να δούμε τι μπορούμε να κινητοποιήσουμε από τα συνταξιδοτικά ταμεία, τα κονδύλια, δηλαδή τα, λεφτά που υπάρχουν αποθηκευμένα στα, στα συνταξιδοτικά ταμεία. Υπάρχουν κλειδωμένα 35 τρισεκατομμύρια ε, δολάρια. Ε, πώς μπορούμε να τα αποδεσμεύσουμε αυτά κάνουμε αυτέ τι συζητήσει. Πολλέ από αυτέ τι συζητήσει έχουν γίνει. Χρηματοδότηση μπορεί να βρεθεί, ε, παραδείγματος χάρη για τη βιώσιμη ενέργεια για όλου. Ε, όταν κοιτάμε τον, τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να βρούμε τα εργαλεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο και να δώσουμε κίνητρα. Αλλά θα πρέπει βεβαίω και οι χώρε να βοηθήσουν, τόσο ώστε να έχουν το κατάλληλο περιβάλλον και να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά ε, γίνεται μεγάλη συζήτηση και για άλλου τύπου χρηματοδότηση. Αλλά ελπίζω στις διαπραγματεύσεις ε, να δούμε ότι οι χώρε ε, δεν θέλουν να χάσουν την. Θα το δείτε, δεν θέλουν να χάσουν την βοήθεια. Θέλουν όλα αυτά τα κονδύλια και όλη αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση να είναι επιπλέον πραγματικά. Πρέπει να έχουμε τη θέληση για να βρούμε, ας πούμε, το, το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε αυτά τα λεφτά για το τρόπο ζωή. Ε, κάνουμε μεγάλη συζήτηση για την εναλλακτική στο σημερινό τρόπο ζωή. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, γιατί όταν κοιτάτε ας πούμε, τις φιλοδοξίες που έχουν οι αναπτυσσόμενοι, ας πούμε, θέλουν να ζήσουν όπως οι βόρειες χώρες, ε, οι χώρες του πρώτου κόσμου. Ε, και πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ ε, λύσεις, ειδικά να προτείνουμε πράγματα στους νέους, γιατί ε, εάν δεν τους πείσουμε για διαφορετικό lifestyle, για διαφορετικό τρόπο ζωής, δεν είναι βιώσιμη αυτή η στόχη. Ε, Επίση, οι επιχειρήσει μπορούν να παίξουν ρόλο εδώ και πρέπει να αντιμετωπίσουν βέβαια και τα αιτήματα των αγορών. Ε, το θέμα, αυτό που είπατε για τους, ε, τη δίωξη των χριστιανών, ε, δεν είναι μόνο θέμα δίωξη ε, χριστιανών. Και διώκονται και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι. Το θέμα είναι οι άνθρωποι, διώκονται άνθρωποι. Ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους καταπατούνται. Δεν πρέπει να ανεχτούμε κάτι τέτοιο. Το να εστιάζουμε στου μένες στου δε, ε, αποκλείουμε τους άλλους. έτσι. Το βασικό είναι ότι όλοι έχουν ε, δικαίωμα στη ζωή και δεν πρέπει να διώκονται φυσικά. Ε, τα έξι στοιχεία. Ε, σίγουρα έχουν μπει στο αρχικό σχέδιο. Είναι τα 5 P τα οποία λέμε, από τα αγγλικά βέβαια. Ο όρος ε, checklist δεν είναι σωστός, λίστα ας πούμε. Αλλά δεν πρέπει να επιτάσσουμε αυτά θα κάνετε στις χώρες. Ε, θα πρέπει απλώς να τι εντάξουμε στις, στην προσπάθεια ε, και να βάλουν την ανάπτυξη στις πολιτικές τους. Ε, με τις επιταγές δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται να προωθήσουμε τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχου με την επιταγή. Θα πρέπει σε επίπεδο χώρα να αναθεωρηθούν τα σχέδια και οι πολιτικές, ώστε να πάνε λίγο παραπέρα και να ενσωματώσουν και την βιώσιμη διάσταση. Ευχαριστούμε. Κλάου δύο λεπτά κανονικά έπρεπε να έχει ο καθένας. Εσείς δύο λεπτά μπορείτε να μας απαντήσετε σε δύο λεπτά. Ναι, θα προσπαθήσω. Την αμήνα έτσι κι και αύριο θα την ξαναδούμε. Έφυγε βέβαια κύριος Βέλε, εγώ δεν θέλω όμως να αποφύγω την ερώτηση που κάνετε. Θα θέλαμε καλύτερο αποτέλεσμα βέβαια και η Επιτροπή το ξέρετε και από τις ανακοινώσεις μας αυτό. Από τη συζήτηση πάντως στο Συμβούλιο καταλήξαμε σε κάτι καλό, γιατί υπήρξε μεγάλη πίεση από πολλές χώρες μέλη για δέσμευση. Και ακόμα αν δεν είναι αρκετά καλό για την Αντισαμπέμπα και άλλες χώρες είπανε να μην υποσχεθούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να τηρήσουμε γιατί διακυδεύεται η αξιοπιστία μας. Οπότε έχουμε ένα συμβασμό. Καλό ή κακό δεν ξέρω, 28 χώρες μέλη πάντως συμφώνησαν και κάποιες από αυτές δεν ε, ξέρουν από αποφάσεις στον τομέα της ανάπτυξης. Συνεπώς πρέπει να δείτε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι αξιοπρεπή συμβασμό αυτός και μας ε, κάνει να λέμε ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα φτάσουμε και νωρίτερα το 0,7% και αποφασίσαμε να στοχεύσουμε και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό, αλλά είναι ένας συμβιβασμός. Ερχόμαστε με μια δέσμευση, άλλοι όχι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε περήφανοι και να το γνωστοποιούμε αυτό. Πράγματι, μερικές φορές δεν τη δείτε. Τώρα, για τα άλλα θέματα. Έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Το εμπορικό καθεστώ μα. Είμαστε η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά, η πιο ανοιχτή στον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Μην το ξεχνάμε. Επίση, εμεί καταπολεμούμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ότι τα παράνο, το παράνομο εμπόριο. Και θα εξακολουθούμε για την ενέργεια, για το κλίμα. Αυτά που κάνουμε στην Ευρώπη είναι πολύ καλά για την ανάπτυξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί κινητοποιούνται πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλα πράγματα. Δίνουμε όθηση για να κινητοποιούνται και ε, από το εσωτερικό πόροι, με διαφάνεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα και πάλι βοηθούμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να κινητοποιήσουν τους δικούς τους πόρους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ροές. Πώς μπορούμε τώρα να δουλέψουμε με τον ιδιωτικό τομέα. Οι δεσμεύτηκαν ε, οι Ηνωμένε με 20 εκατομμύρια για τις αφρικανικές χώρες. Εμείς θα το κάνουμε αυτό με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας θα μεταφέρει την ενέργεια στους Αφρικανούς με εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, άρα καταπολεμούμε και την κλιματική αλλαγή. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά προγράμματα για να μεταφέρουμε ηλεκτρισμό στην Αφρική, αλλά ο ιδιωτικό τομέας θα δεσμευτεί και θα έχουμε έτσι ένα ιδιωτικό τομέα στην Αφρική και η ενέργεια με, από εναλλακτικέ πηγές θα υπάρχει στην Αφρική. Έτσι θα συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλω να πω κάτι και για την οικουμενικότητα. Έφυγε βέβαια ο κύριος Έικ, αλλά από την ερώτησή του ετέθηκε το θέμα της διατροφής. Μα ακριβώ γι' αυτό η οικουμενικότητα είναι σημαντικό. Πρέπει το θεματολόγιο αυτό να φτάσει στην κοινωνία των πολιτών. Δεν είμαστε εμεί που θα πούμε στον κόσμο πώ θα τρέφεται. Είναι η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτε που θα καταλάβουν ότι πρόκειται για αλλαγέ, ότι αυτό το θεματολόγιο έχει αλλαγέ. Η κοινωνία των πολιτών δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι αλλαγέ αυτέ που θα προκύψουν. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά Θέλω να τηρήσω τι οδηγίε που μου δώσατε και να περιοριστώ στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ κλάου. Μπορούμε έτσι να κλείσουμε το πρώτο μα πάνελ. Έχουμε μια κρίσιμη στιγμή σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει πριν από την Αντίσα Χρειάζεται μια ηγετική θέληση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά. Συγγνώμη για το επόμενο πάνελ λοιπόν και α δώσω το λόγο το νέο ε, διευθύντη τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ αυστηρότερο σε ό,τι αφορά τον χρόνο. Ζητώ συγγνώμη από τους ομιλητές. Λοιπόν, το δεύτερο πάνελ αφορά τις ε, πτυχές του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την ατζέντα της ανάπτυξης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει δύο σημαντικά θέματα που την ενδιαφέρουν, που συνάπτονται ιδιαίτερα με την ατζέντα της ανάπτυξης, η κατάσταση του περιβάλλοντος και τα θέματα κλιματικής αλλαγής και το θέμα των ε, ζητημάτων δημόσιας υγείας. Οι δύο συμμετέχοντες λοιπόν στο πάνελ θα μας δώσουν κάποιες πληροφορίες για την κλιματική πλευρά και την πλευρά βιωσιμότητας της επίτευξης των στόχων σε αυτό το, χώρο και θα μας δώσουν περισσότερες ε, λεπτομέρειες για τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή εστίασης από μια προοπτική απλώς ανάπτυξη σε μια προοπτική βιώσιμη ανάπτυξη. Η κατάσταση του περιβάλλοντος εδώ πέρα είναι πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ανάπτυξη και δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της ανθρώπινης ανάπτυξης χωρίς να συζητήσουμε το θέμα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Γι' αυτό συμφωνώ λοιπόν με όλους αυτούς οι οποίοι διεκδικούν πρόσθετες ε, συμμετοχές επιτροπών σε αυτήν τη συνεδρίαση. Οι δυο μας επιτροπές όμως, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή για την Ανάπτυξη νομίζω ότι συμφώνησαν να έχουν αυτή την κοινή συζήτηση στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στους δύο ομιλητές σε αυτό το πάνελ καταρχήν τον κύριο Ρομπέρτο Μπερτολίνη, ο οποίος είναι, ε, είναι κύριος ε, επιστήμων και εκπρόσωπος του Οργανισμού για την ε, ε Παγκόσμιο Οργανισμό για και τον κύριο Ζάνος Σλίνσκι, ο οποίος είναι Διευθυντής της Ακαδημίας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεν θα στο περισσότερο χρόνο, ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε λίγο από τον χαμένο χρόνο τον οποίο αναζητούμε και να μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε και πάλι το χρονοδιαγραμμά μας και να τον λόγο στον κύριο Μπερτολίνη. Σε ευχαριστώ κύριε Γιάβορ, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επιτροπή Περιβάλλοντος που με προσκάλεσε να σας παρουσιάσω αυτά τα οποία πιστεύουμε γιατί νομίζουμε ότι η προστασία και η πρόθεση της υγείας είναι ένας κύριος συντελεστής στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων. Θα είμαι λίγο πιο τεχνικός από ότι στις προηγούμενες συζητήσεις, αλλά είναι χρήσιμο να μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις για να καταλάβουμε καλύτερα πώς συνδέονται οι διάφοροι παράγοντες σε επόμενη διαφάνεια. Τα τελευταία χρόνια η υγεία έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, οικονομικό θέμα και θέμα ασφάλειας, ένα κοινωνικό αγαθό, ένα συλλογικό αγαθό για το οποίο χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Είναι Μεγάλη η επένδυση λοιπόν που απαιτείται στον τομέα αυτό είναι ένα σημαντικό οικονομικό τομέα και ένα τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνική δικαιοσύνη. Μία από τι κύριε μελέτε που έχει διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ ανάπτυξη και υγεία, υγεία και ανάπτυξη, δημιουργήθηκε από την Επιτροπή για την Υγεία στι αρχέ του 21ου αιώνα και τόνισε πώ μπορεί η υγεία να συμβάλλει στην πολιτική ατζέντα ανάπτυξης. Ίσως δεν μπορείτε να δείτε πολύ καλά τι λέει αυτό το γράφημα στο πίσω μέρος της έσως, αλλά λέει ότι η επιρροή της ε, υγείας σε, μακρο, σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, την παιδεία κτλ. Και η ανάπτυξη μαζί με τη μείωση της ένδυας έχουν σημαντικό χαρακτήρα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό γιατί αναφέρθηκε για το θέμα των δικτών πρέπει <clears throat> να βρούμε σε ορισμένου δείκτε οι οποίοι κάπω θα μπορέσουν να συνοψίσουν τι διάφορε πτυχέ τη ανάπτυξη και η υγεία ίσω είναι ένα από αυτά. Η επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ πάλι είναι αόρατο αυτό το γράφημα από το πίσω μέρος αίθουσας, αλλά βλέπετε εδώ την σύνδεση μεταξύ προσδοκίμου ζωής και κατακεφαλήν ΑΕΠ. Βλέπετε ότι το αυξανόμενο κατά κεφαλή ΑΕΠ οδηγεί σε μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωση. Ενώ η μείωση του κατακεφαλήν ΑΕΠ οφείλεται και σε ανισότητες και ελλείψεις στο σύστημα διανομής στις χώρες που έχουν προβλήματα. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν με την ατζέντα των βιώσιμων στόχων είναι να μειώσουμε τις ε, ανισότητες και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του υγειονομικού συστήματος από την άλλη πλευρά. Η υγεία έχει σημαντική ανάπτυξη. Ακεί επιρροή, παραγωγός χάρη, η απουσία από τη δουλειά λόγω ασθένειας ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο περίπου 2,5% του ΕΠ και επίσης επηρεάζει την, ε, το προσδόκιμο επιβίωση. 1% σε, στο προσδόκιμο επιβίωση σημαίνει 6% αύξηση στο ΑΕΠ και 10% μείωση ε, τα προβλήματα υγείας οδηγεί σε ανάπτυξη του ΑΕΠ. Οι στόχοι λοιπόν αυτοί που θα αντιμετωπιστούν στην ε, συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας περιλαμβάνουν και το θέμα της υγείας ως στόχος 3 με μια δήλωση υψηλού επίπεδου για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το υγιεινό τρόπο ζωής σε όλες τις ηλικίε. Με τους 13 επιμέρους στόχους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε ασθένειες και τους παράγοντες που τις ενισχύουν. Να σας δω τώρα για ορισμένου στόχους. Για τον τρίτο στόχο βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πρώτοι στόχοι αντιμετωπίζουν πράγματι θέματα που ήταν τμήματα των στόχων της χιλιετίας. που απαιτούν περαιτέρω προσπάθεια για να μπορέσουν να εδραιωθούν οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα. Παραδείγματο να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα, να μειωθούν οι θάνατοι των νεογνών και των ε, βρεφών, να αντιμετωπιστεί η επιδημία του AIDS της ε, θυματίωσης κτλ. Αλλά θέλω να δώσω περισσότερη έμφαση σε ένα στόχο που αφορά τις μη μολυσματικές ασθένειες για ένα συγκεκριμένο λόγο. Στον κόσμο αντιμετωπίζουμε τώρα μια μεγάλη επιδημιολογική μετάβαση. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι μολυσματικές ασθένειες δεν είναι πια ο κύριος λόγος θνησιμότητας. <clears throat> Και αυτό τροποποιεί κατά ανάγκη την ε, αντιμετώπιση την αναπτυξιακή που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις μολυσματικές ασθένειες και την υγεία των λεχονών και των βρεφών. Φυσικά πρέπει να συνεχιστούν να υποστηρίζονται αυτή οι στόχοι, αλλά πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο στις προσθετες προκλησει προκλήσεις. 50-70% των φτωχών ζουν τώρα σε χώρε μέσου εισοδήματο και η οικονομική ανάπτυξη και ο συγχρονισμό έχουν βελτιώσει, έχουν οδηγήσει στη δυνατότητα να υπάρχει μια μορφή υγεία η οποία δεν είναι υγιεινή. Και υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνο αυτός. Οι αναπτυσσόμενε χώρε λοιπόν αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι προβλήματα αναπτυγμένων χωρών. Όλο και περισσότερο το βάρο πέφτει σε χώρε, οι οποίε είναι ενδιάμεσε, όπου τα άτομα αναπτύσσουν ασθένειες νωρίτερα από ότι ε, στις πλούσιες χώρες. Ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μόνο οι ασθενείς, μόνο οι γέροι και οι ασθενείς μπορούν να πεθαίνουν. 12 εκατομμύρια πρόορη θάνατοι το χρόνο δημιουργούνται το, από μη μολυσματικές ασθένειες. Σε ορισμένε αναπτυσσόμενες χώρε τη Ασία, ο αριθμό των θανάτων από καρδιοαγγειακές ασθένειες πριν από τα 55 πλησιάζει τον, το, αυτών των αναπτυγμένων χωρών. Η, η διεθνή κοινότητα έχει κάποια εργαλεία για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό η δήλωση του 2011 για τις μη μεσοματικές ασθένειες δίνει κάποιες τέτοιους δρόμους. Η Γενική Συνέλευση του 2014 στα Ηνωμένα Έθνη είδε ότι δεν υπήρξε έλλειψη πολιτικής θέσμευσης, αλλά έλλειψη ικανότητας να δράσουμε λόγω έλλειψης εθνικής εμπειρογνωμοσύνης σε χώρες με μέσο και χαμηλό εισόδημα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη συνεργασία για να δοθούν μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη στο μέλλον. Για τους στόχους λοιπόν που αναφέραμε θα ήθελα να υπογραμμίζω και μια άλλη πτυχή ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ της ένδυας και των μη μολυσματικών ασθενειών αλλά πρέπει να δούμε τους τρόπους να αυξήσουμε την πρόσβαση στην ε, περίθαλψη και να μειώσουμε και το κόστος της περίθαλψης που στέλνει πολλές οικογένειες κάτω από την γραμμή ένδυας. Η παγκόσμια, η οικουμενική, η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους στόχους μας. Η δήλωση των ΗΠΑ τονίζει την ανάγκη να υπάρξει τέτοια οικουμενική κάλυψη για να φτάσουμε τους στόχους της χιλιετίας. Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει δείχνουν ότι οι καταστροφικές δαπάνες έχουν οδηγήσει 150 εκατομμύρια άτομα κάτω από την γραμμή ενδίας. Και αυτό κάθε χρόνο. Ενώ πολλές κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να αφήνουν τους ανθρώπους κάτω από τη γραμμή της ένδυας, αλλά αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια πηγή περαιτέρω ένδυας. Πρέπει αυτή η διαδικασία να λειτουργήσει σε επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα και τους θεσμούς κάθε χώρας, την ιστορία των υγειονομικών του συστημάτων και τις προστοκίες των πολιτών. Μετά από δεκαετίες εμπειρίας, ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν θα γίνει ένας δίκαιος χώρος υγειονομικής περίθαλψης από μόνος του. Το σύστημα δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισότητα, ή προς παγκοσμία κάλυψη. Οι οικονομικές αποφάσεις μέσα σε κάθε χώρα δεν οδηγούν αυτόματα στην προστασία των φτωχών και την πρόωθηση της υγείας τους. Οι παγκοσμιοποίηση δεν είναι αυτορυθμιζόμενη προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, αν αυτών, δεν θα οδηγήσουν σε υγειονομική ισότητα ή σε πρόσβαση στην υγεία για όλους. Όλα αυτά απαιτούν μια θεληματική πολιτική και μόνο με αυτή την οικονομική προσέγγιση μπορούμε να έχουμε πρόθεση της ανθρώπινης υγείας και ανάπτυξης. Μόλον τούτο, όπως ελέγχθηκε στη συζήτηση, μέσα από μια προοπτική βιώσιμη ανάπτυξη, η υγεία συνδέεται με άλλους στόχους της ε, ανάπτυξης, βιώσιμους στόχους. Επηρεάζει τα θέματα της ε, υγείας, της ε, γεωργίας, της ποιότητας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύπλοκη αυτή, αυτή η διαφάνεια και δεν μπορώ να την αναλύσω πλήρως. Αλλά αντιμετωπίζει μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και η οποία νομίζω θα καλυφθεί και στην επόμενη παρουσίαση που είναι η κλιματική αλλαγή. Όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής μας, είναι το ουσιαστικό θέμα σε επίπεδο πολιτικής του 21ου αιώνα. Όπως φαίνεται σε αυτές τις διαφάνειες, οι κλιματικές ε, συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και να δημιουργήσουν μηχανισμούς που ευνοούν μεγαλύτερη ε, επιπολασιμότητα των ασθενειών λόγω μεγαλύτερης υγρασία ή άλλων συνδικών προστασία λοιπόν τη υγεία σημαίνει θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υγεία στου διάφορου τομεί όπω ελέγχθηκε προηγουμένω. Η επόμενη διαφάνεια. Εν κατακίνηρη. Η υγεία είναι μια σημαντική συνιστόσα τη υγεια σημαινει θα πρεπει να αντιμετωπισουμε την υγεια στου διαφορου τομει οπω ελεγχθηκε προηγουμενω η επομενη διαφανεια εν η υγεια ειναι μια σημαντικη συνιστοσα της ανθρωπινης ανάπτυξης και της ευμάρης και μπορεί να συμβάλλει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο στόχος της υγείας θα πρέπει να είναι να βελτιώσει την υγεία σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Αυτό σημαίνει να επιταχύνουμε και να συμπληρώσουμε το έργο για τους στόχους της χιλιετίας και να προχωρήσουμε να συμπεριλάβουμε και τις μη μολυσματικές ασθένειες. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις θα τεθεί ένα αμφιβόλο η βιώσιμη ανάπτυξη. Να κλείσω με τα λόγια της Γενικής Διευθύντριάς μας, η οποία πρόσφατα ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε ότι η υγεία είναι κάτι που πρέπει να είναι υποχρεωτικό στοιχείο οποιασδήποτε ατζέντα μετά από το 2015 και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόοδο στην ε, εξάλληψη της ένδυας και της ανισότητας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννο Σλίνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω και να μιλήσω στο αξιότιμο αυτό ακροατήριο. Θα σταθώ μόνο σε κάποιες διαφάνειες. Την παρουσίαση νομίζω θα την έχετε θα είναι διαθέσιμη για εσάς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η διαφάνεια αυτή έχει μία δήλωση ε, μετά από μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge πριν από 12 χρόνια. Οι ερευνητές, επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην διάσκεψη, μάλλον στην έρευνα αυτή, μιλούν εκ μέρους του αυτού τους. Θέλω να πω, δεν μιλούν εκ μέρους των επιχειρήσεών τους, μιλούν προσωπικά, δίνουν την προσωπική τους άποψη. Και από την έρευνα αυτή, το βασικό ερώτημα ήταν, το πρώτο μάλλον ερώτημα ήταν ποιος είναι ο βασικός ο στόχος μιας καλής οικονομίας. Και όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, τα πολλά από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους συμπεριλαμβάνονται και εδώ. Δηλαδή η βελτίωση της ευημερία όλων των ανθρώπων, των μελλοντικών γενναίων επίσης, ισότητα, να λάβουμε υπόψη μας ε, τους περιορισμούς της φύσης και ε, συμμετοχή όλων. Επόμενη διαφάνεια εδώ. Βλέπετε το σχήμα αυτό είναι ένα ντόνατ, το οποίο προσπαθεί να βάλει τους διάφορους παράγοντες στο σχέδιο αυτό. Πρόκειται για την εξή έννοια, ότι η ανθρωπότητα και η κατάσταση στην οποία ζούμε πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν μπορεί να πάμε πέρα από αυτό το lifestyle μας δεν μπορεί να ξεπερνάει κάποιους περιορισμούς που μας βάζει η φύση και ο πλανήτης. Και από την άλλη μεριά η ανθρώπινη κατάστασή μας δεν μπορεί να πάει κάτω από κάποια όρια. Στόχος λοιπόν της εφαρμογής των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων είναι ακριβώς τα έθνη και ανθρωπότητα να βρεθούν μέσα σε αυτό το μεσαίο κομμάτι το πράσινο. Κυρίε και κύριοι πρέπει να σας πω ότι καθώς μιλάμε δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη αυτό που να μπορεί να βρίσκεται στο πράσινο αυτό τμήμα. Είτε βρίσκονται στο μεσαίο κύκλο, δεν έχουν αρκετά ανθρώπινα δικαιώματα, η ανθρώπινη εξωπρέπεια ή από την άλλη μεριά βρίσκονται εκτός με υπερβολικό, υπερβολικά υλικά αγαθά και μη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται και ο τίτλος αυτού του τμήματος εδώ που συζητάμε είναι γιατί χρειαζόμαστε σαφείς βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Γιατί χρειαζόμαστε ταυτόχρονα αυτούς τους στόχους, δηλαδή και κλιματική αλλαγή να αντιμετωπιστεί και προσθέσεις του περιβάλλοντος και υγεία και οικονομία και οτιδήποτε άλλο. Γιατί, γιατί το σύστημα στο οποίο ζούμε είναι ένα περίπλοκο και ήρθε η ώρα να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αλλά μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτό το ερώτημα γιατί έχουμε αυτούς τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Προχωράμε στις διαφάνειες για να προλάβουμε. Γιατί, γιατί είναι επικίνδυνη η κλιματική αλλαγή, γιατί, γιατί, γιατί, υπάρχουν εδώ τα διάφορα ερωτήματα και φτάνουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Το ερώτημα είναι τους χρειαζόμαστε όλους, είναι όλοι εντάξει, τι γνώμη πρέπει να έχουμε για αυτούς και πώς θα τους εφαρμόσουμε. Πώς ξεπερνάμε την κακοφωνία μιας ορχήστρας όταν δοκιμάζει τα όργανα πριν περάσει στην συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε τους στόχους αυτούς, είναι 17, να τους δούμε στο διαδίκτυο, να τους μελετήσουμε, είναι συνολική, είναι πλήρης. Πρόκειται για το θεματολόγιο, το θεματολόγιο. Και πρέπει να σας πω αν θέλετε τη γνώμη μου ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία βασικά που έχουμε να δημιουργήσουμε έναν δίκαιο και ευημερούντα κόσμο για τους αυτούς μας. Τώρα ανάμεσα σε αυτούς τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους υπάρχει και ένας για την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για το στόχο 13. Ελπίζω να είναι τυχερό νούμερο αυτό το 13 που λέει ότι πρέπει να λάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Και είναι ο μόνος που εμφανίζεται με αστερίσκο. Και γιατί, γιατί κάνει μνήμα στις συζητήσεις που θα γίνουν στο Παρίσι των Ηνωμένων Εθνών, του UNFCCC, και μπορούμε έτσι να έχουμε συγκεκριμένα και ποσοτικά εκφρασμένα μέτρα προς τα τέλη της χρονιάς που να τα δεχτεί η διεθνής κοινότητα στο Παρίσι. Είναι λοιπόν ο μόνος στόχος που παραμένει ανοιχτός. Αν το κοιτάξουμε όμως λεπτομερέστερα τον στόχο αυτό θα δείτε ότι ο στόχος αυτός περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Δεν είναι όμως, δεν είναι όμως τα μόνα μέτρα, οι μόνοι στόχοι αυτοί οι πέντε που βλέπετε εδώ. Αν τους κοιτάξετε πιο συγκεκριμένα, θα δείτε ότι όντως μπορούν να βοηθήσουν, αλλά προχωρώντας πιο πέρα καταλαβαίνουμε ότι σε ένα περίπλακο σύστημα μια κάθετη προσέγγιση μονομερής δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ας πάμε πιο πέρα και πιο πέρα. Να, αυτό είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε σήμερα, στην πραγματικότητα. Είναι ένα σύστημα φύσης κοινωνικό, οικονομικό. Είναι ένα σύστημα όμως σαν μια ματριόσκα, δηλαδή με τις κούκλες που μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Υπάρχει φύση, μέσα έχουμε την κοινωνία και πιο μέσα έχουμε την οικονομία. Σας λέω ίσως τα προφανή. Αλλά αν δείτε η, τα συνήθεια βιβλία για την οικονομία δεν παρουσιάζουν έτσι την οικονομία. Θα δείτε τον κύκλο φύση σαν ένα πολύ πολύ μικρό κομματάκι που να εξαρτάται από την οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει μια ιεράρχηση, ότι το σύστημά μας είναι ιεραρχημένο. Ένα σύστημα είναι ο μεγάλος κύκλος, μέσα ένας πιο μικρός και ένας πιο μικρός. Υπάρχουν ε, και διάφορα υποσυστήματα βέβαια που έχουν να κάνουν με τη τεχνολογία, με τις αξίες, με το κεφάλαιο, με την τροπή κλπ. κλπ. Αν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό ακριβώς είναι που έχουμε στο σύστημά μας. Η κλιματική αλλαγή λαμβάνεται υπόψη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι στόχοι που βλέπετε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, έχουν να κάνουν με την ε, υγεία, τις φυσικές καταστροφές που πρέπει να περιοριστούν. Εδώ βλέπετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πώς μετρούνται, πώς ε, και πού δημιουργούνται στη βιομηχανία, στο δρόμο, στις πόλεις μας κλπ. κλπ, στη γεωργία, έτσι. Τέλος, Η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση της έχει να κάνει βέβαια με τη φύση. Η φύση βοηθάει για να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τους ωκεανούς, για τη χρήση γης, για την βιοπικιλότητα, για τα δάση. Πρόκειται για να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και η ζωή μας να γίνεται πιο καθαρή και να συνάδει καλύτερα με τους πόρους αυτούς. Τότε θα προστατευτούμε. Και έτσι φτάνουμε στους στόχους πέντε συν που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αν όμως κάνουμε το ίδιο και για την υγεία ή αν κάνουμε το ίδιο για τα δύο φύλλα, αν κάνουμε το ίδιο για τη βιοπικιλότητα, θα μπορούσα να κάνω το ίδιο ακριβώς για όλους αυτούς τους στόχους, ότι δηλαδή πέρα από τους στάνταρ στόχους για όλα αυτά τα θέματα, για το νερό για παράδειγμα, στις άλλες στήλες περιλαμβάνονται μέτρα και στόχοι οι οποίοι λειτουργούν για το συγκεκριμένο στόχο. Καλά. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τους στόχους και τα μέτρα που παίρνουμε. Αυτό το 5 24 δείχνει πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα και πώς το ένα πράγμα μπορεί να επηρεάζει το άλλο, πώς όλα είναι αλληλένδετα και πώς το ένα μπορεί να μετριάζει τα αποτελέσματα του άλλου ή αντίθετα να τα ενισχύει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό το μοντέλο. Και επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω. Αν δείτε την μελέτη πώς το σημερινό σύστημα λειτουργεί των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και κατά πόσο βοηθάει αυτό εδώ το σχήμα, το donut που σας έχω ζωγραφίσει εδώ, Δεν είναι κάτι που έχω κάνει εγώ. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το έκανε, έτσι. Βρήκαν ότι οι στόχοι και τα μέτρα, εφόσον εφαρμοστούν, μπορούν να μας βάλουν και πάλι όλους, από όπου και αν προερχόμαστε, είτε εκτός των κύκλων, είτε στο μέσα κύκλο. Αξίζει να το δοκιμάσει κανείς. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε αυτό το πολλά υποσχόμενα σχέδιο για το μέλλον είναι μια μοναδική διαδικασία. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες. Καταλήξαμε σε αυτό μετά από τη διαβούλευση που είχαμε την επιστημονική κοινότητα με πολιτικούς και λαμβάνοντας υπόψη μας συγκεκριμένα στοιχεία. Και ξέρουμε τι θα γίνει αν συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, business as usual. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική και σας ευχαριστώ όλες τις χώρες μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκ μέρους των συμπροέδρων, αν μπορώ να το πω έτσι. Περάστε στην εφαρμογή όμως. Ίσως να είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ οι βουλευτέ. Μήπω έχουν ερωτήσει τώρα. Κυρία Βεσέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντες οι δύο μιλητές. Για τον κύριο Μπερτολίνη μία ερώτηση που μίλησε στους βασικούς στόχους ε, της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης. Ε, δικαιοσύνη και δικαίωμα στην υγεία. Ε, χρειάζεται επιχρηματοδότηση για πρόσβαση στα βασικά φάρμακα. Ποια είναι η γνώμη σας για την αίτηση του Μπαγκλαντές το Φεβρουάριο ε, στη χώρα των λιγότερων εμπτυγμένων χωρών για μια επέκταση στη μεταβατική περίοδο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των διαφορών χωρών σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ο ΙΕ είπε ότι οι χώρες αυτές επηρεάζονται αρνητικά, ειδικά ε, από τα TRIPS ε, για τα φάρμακα και τα ιατρικά προϊόντα. Να σας ρωτήσω κύριε Μπερτολίνη, αν συμφωνείτε με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη να επεκταθούν αυτές οι εξαιρέσεις για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και αν ναι, Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι πρέπει να επεκταθεί αυτή, να παραταθεί αυτή η εξαίρεση, ούτω ώστε να υλοποιήσουμε του στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω κάτι να ρωτήσω τον κύριο Περτολίνη. Και το TTIP. Συμφωνείτε τη στιγμή που έχει να κάνει με το εμπόριο, με συμφωνίες. Ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα υγείας, αλλά και όχι μόνο. Οπότε ποια είναι η άποψή σας για την συμφωνία αυτή που συζητάμε. Δεύτερον, μιλάμε για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Η δικιά μου χώρα παρακολουθεί αυτό το θέμα πολύ. Η... Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα, γιατί η Κίνα δεν έχει κάνει τίποτα. Μπορείτε να πείτε η Ευρώπη τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε. Κύριε Χαβέρ. Ευχαριστώ πολύ για τις δύο αυτές τόσο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Κύριε Περτολίνη, δείξατε τη σύνδεση μεταξύ οικονομίας και ένδυας και υγιές. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται πάντα σε όλες τις μελέτες, αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά δεν, εξασ... δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το συντονισμό της παροχής υγειονομικής περίθαλψης ώστε να καλύπτει όλους τους ανθρώπους τη αναπτυσσόμενη χώρες. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά το θέμα αυτό για μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα κύριε Σελίνσκι. Επίσης και αυτό που είπατε ήταν ιδιαίτερα, αυτά που είπατε ήταν συναρπαστικά αλλά έχω την εντύπωση ότι από τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης έχουμε λάβει πολύ περιορισμένα υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Είπατε ότι κάποια πράγματα παραμένουν ανοιχτά και περιμένετε τη διάσκεψη του ε, Παρισιού. Μήπως θα πρέπει και ο στόχος του να μην ξεπεράσουμε το, τους δύο βαθμούς ε, αύξηση θερμοκρασία του πλανήτη να λυθεί υπόψη. Και επίσης μιλήσατε για τα πλανητικά όρια και δείξατε τους τρεις κύκλους που δείχνουν γιατί τα όρια του πλανήτη θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα οριακών συνθηκών. Και αν δεν βάζετε την οικονομία <clears throat> στο κέντρο, αλλά τον άνθρωπο ως μέτρο των πραγμάτων μέσα σε αυτή την πλανητική απεικόνηση, θα ήταν ίσως καλύτερο έχετε δείξει στις άλλες σας τις διαφάνειες πόσο μεγάλη η ανισότητα που μπορεί να υπάρξει. Ίσως όταν ο άνθρωπος μπει στο κέντρο να αυξηθεί και η ισότητα. Thank you. And I would like to give the floor to our speakers. To... Τώρα θα απαντήσουν οι ομιλητές μας. Ο κ. Περτολίνη πρώτος. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσες, όντως. Συμφωνώ με τη θέση που έχουν κάποιες υπηρεσίες του ΟΗΕ ότι η παράταση της άδεια άνευ περιορισμών θα πρέπει να δοθεί σε αυτές τις χώρες. Αν θέλουμε, από τη μία θέλουμε να καλύψουμε όλους ε, με υγειονομική περίθαλψη δηλαδή και από την άλλη να προστατεύσουμε πολλούς ανθρώπους ε, από διάφορες ασθένειες λόγω φτώχειας. Αν θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε την καθολική υγειονομική περίθαλψη, αυτό πρέπει να το κάνουμε πρέπει να παρατείνουμε αυτή την άδεια. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι σημαντικό να παραταθούν αυτέ τι συμφωνίες, γιατί αλλιώς ε, θα έχουμε μείζωνα προβλήματα σε κάποιες από αυτές τις χώρε χαμηλού εισοδήματο. Ε, τώρα, σε σχέση με το TTIP. Ε, η ανησυχία μας στον ΠΟΗ αφορά περισσότερο τα εξή θέματα. Όταν μιλάμε για αυτή την συμφωνία τύπου. φυσικά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι θα εμπεριέχει. Το βασικό πρόβλημα είναι να εξασφαλίσουμε ότι πολλά από τα στοιχεία πρόοδου που έχουμε στην Ευρώπη, στο κανονιστικό επίπεδο, ε, στα χημικά, στον έλεγχο της έκθεσης απέναντι σε διάφορες ουσίες, όλα αυτά να μην παραβιαστούν, να μην εγκαταληφθούν λόγω αυτής της νέας συμφωνίας. Τι τύπου. Η προσπάθεια που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος να μην διακυβευτεί λόγω αυτής της εμπορικής συμφωνίας. Υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα στις πολιτείες γιατί δεν προστατεύουν την ε, υγεία και το περιβάλλον όπως εμείς. Μπορούμε να δούμε τις στατιστικές. Δεν είναι περίεργο. Βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο, στην κατάσταση της υγείας των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην παραιτηθούμε από, τις, από τα μείζωνα επιτεύγματά μας στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την μικροβιακή αντίσταση, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί η Κίνα στην τελευταία συνάντηση στη Γενέβη ε, το Μάιο, μαζί με διάφορες άλλες χώρες, ε, προσυπέγραψε ένα μεγάλο ψήφισμα για ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατά της ε, μικροβιακής αντίστασης. Άρα μάλλον και οι Κινέζοι ξέρουν αυτό το πρόβλημα. Ίσως ε, δεν είναι δεν γνωστό αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει στην ατζέντα και για πρώτη φορά έχουμε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και τώρα υπάρχει κίνδυνο στο μέλλον να μην έχουμε αρκετά αντιβιωτικά για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ε, τις κλασικές τρέχουσες ασθένειες. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε, να ρυθμίσουμε την ε, χρήση των αντιβιωτικών, αλλά να προωθήσουμε και την έρευνα στον τομέα αυτό. Και η Κίνα είναι και αυτή εταίρος όλη την προσπάθεια αυτή. Ενέκρινε αυτή την συμφωνία, όλοι την ενέκριναν. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας. Είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντίστασης. Σε ό,τι αφορά την καθολική υγειονομική περίθαλψη και την πρόσβαση στα φάρμακα. Προσπάθησα να σας δείξω ότι αυτή η περίθαλψη είναι βασικό στοιχείο, είναι βασική προϋπόθεση αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος που έγινε στο επίπεδο της ευημερίας σε πολλές χώρες εξακολουθεί να υπάρχει και απέναντι στις ασθένειες και στην αναπηρία. Πολλοί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χάνουν πόρους αφαιρούνται από τη διατροφή τους, την εκπαίδευσή τους, από την ευμερία των παιδιών τους, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως έδειξαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τις διάφορες πτυχές. Οι περισσότερες από αυτές τις πτυχές για τις οποίες μιλάμε είναι αλληλένδετες και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν και κάποια ερωτήματα. Ναι, αν μπορώ να γυρίσω πίσω σε κάποιες διαφάνειες. Η κλιματική διάσταση πρέπει να συμπεριληφθεί στην ε, προβληματική μας για το θέμα των δύο βαθμών και τη μη υπέρβαση των δύο βαθμών σαν όριο. Έχουμε ένα πρόημιο βέβαια πολύ σημαντικό στο έγγραφο που πρέπει να το μελετήσουμε και θα πρέπει να εργαστούμε με αυτό και να δημιουργήσουμε ένα κοινό, ε, μια κοινή ονοματολογία. Νομίζω ότι κατανοίγουμε σε μια κοινή συναντήληψη για όλα αυτά. Στο προήμιο αυτό, όχι μόνο οι δύο βαθμοί, αλλά και ο στόχος της μη υπέρβασης των 1,5 βαθμών αναφέρεται και υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές συμφωνίες σε επίπεδο πολιτικό. Αναφέρονται ως βάσεις για, τα, για τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε και περισσότερο. Αν αυτοί οι στόχοι λοιπόν που αναφέρονται για την επίτευξη δέσμευσης άνθρακα αν μπορούν να εφαρμοστούν θα είμαστε ασφαλείς. Και ένα από τα θέματα αυτά είναι η αύξηση του pH των ε, ωκεανών, της ε, οξύτως μάλλον των ε, ωκεανών. Δεν αρκεί λοιπόν να μην έχουμε περισσότερο διοξίδιο άνθρωπο στην ατμόσφαιρα, θα πρέπει να σταματήσουμε και την αύξηση τη οξύτητα των ωκεανών και αυτό σημαίνει πρέπει να σταματήσουμε τις εκπομπές αριών θερμοκηπίων. Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε από όλες τις πλευρές, δεν μπορούμε να καλύψουμε μονάχα ένα τμήμα του προβλήματος, αλλά όλες τις πλευρές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορέσουμε να πετύχουμε να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς και να γυρίσω περισσότερο μία ακόμα α, εδώ πέρα με τον άνθρωπο στο κέντρο. Είναι ερετικό ίσως. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν το να δεχτούν ότι το πλανητικό σύστημα είναι κλειστό, είναι πεπερασμένο. Οι μικρότεροι κύκλοι μπορούν να, βγουν, να αυξηθούν και να αναπτυχθούν μόνο σε βάρος της ε, φύσης. Είναι σύστημα μηδενικού αθροίσματος. Η ανθρωπότητα λοιπόν επεκτείνεται σε βάρος της φύσης. Αυτό είναι δεδομένο. Και η οικονομική ανάπτυξη είναι υποσύστημα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν είναι όλη η δραστηριότητα της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα δεν είναι υποσύστημα της οικονομίας. Η οικονομία είναι υποσύστημα της ανθρωπότητας. Πρέπει να μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Ότι είναι παίγνιον μηδενικού αθροίσματος και είναι σαφή τα όρια, τα εξωτερικά όρια. Ευχαριστώ. Thank you very much. And, uh, Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές και σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Για να συνοψίσουμε και να τελειώσουμε αυτό το τμήμα της ακρόασης θα επανέλθω σε κάτι που απορρέει από αυτά που είπε ο κύριος Μπερτολίνη για το πώς αναπτύσσεται η οικονομία και πώς τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται προβλήματα φτωχών χωρών, προβλήματα πλουσίων χωρών και για σας κύριε Σλίνσκι θα έλεγα ότι αυτό εδώ το, αυτή η διαφάνεια όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα με τους κύκλους, ομόκεντρους κύκλους αλλάζει τον τρόπο σκέψης μας όσον αφορά την ανάπτυξη. Συνήθως συζητάμε για την ανάπτυξη μιλώντας για κάτι που έχουμε εμείς στις πλούσιες χώρες και που λέμε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να δώσουμε κάτι στις αναπτυσσόμενες χώρες από αυτά που εμείς έχουμε. Αλλά αν λάβουμε υπόψη μας τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι τελώς διαφορετική. Είναι πολλά πράγματα που αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να έχουν και που εμείς δεν έχουμε στον αναπτυγμένο κόσμο. Οι σημεία αναπτυξιακοί στόχοι λοιπόν είναι κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και εμείς έχουμε πολλά να κάνουμε στις πλούσιες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή, για τη βιοποικιλότητα και πολλά άλλα, τους ωκεανούς κλπ. Έτσι η συζήτηση και ο τρόπο σκέψη μα για την ανάπτυξη γίνεται εντελώ διαφορετικό από ό,τι κατά το παρελθόν. Πώ όμω να του εφαρμόσουμε αυτού του βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου, αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στο τρίτο πάνελ. Η Έλλη Σλάιν θα προεδρεύσει. Πρόκειται για την εφαρμογή των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. good afternoon. Γεια σα. Καλώ ήρθατε βέβαια εδώ πέρα. Ε, λέγομαι Έλλη Στάιν. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Ανάπτυξη Στη σοσιαλιστική ομάδα είναι τεράστια η χαρά για μένα να είμαι επικεφαλή του πάνελ αυτού που έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων. Οι προηγούμενοι ομιλητέ έχουν ήδη υπογραμμίσει τη σημασία τη ανάγκη εφαρμογή τεράστια προσπάθεια και πάρα πολλή χρόνο τα πανάτε στο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τη στρατηγική βιώσιμων στόχων αυτό το Σεπτέμβριο. Πέραν όμως από τους στόχους θα πρέπει να δούμε πώς αποτελεσματικά θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους βιώσιμους στόχους ξεκινώντας από την διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην Αντισαμπέδα. Είναι φιλόδοξη η ατζέντα και είναι τεράστιες οι προκλήσεις. Προφανώς τα χρήματα είναι σημαντικά και ο ρόλος του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για χρηματοδότηση είναι σημαντικός. Η κινητοποίηση περαιτέρων πόρων για να συνεχίσουμε τον αγώνα για τους στόχους θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται καλύτερη χρησιμοποίηση των ενδογενών πόρων όπως είπε και η Αμίνα Μοαμέτ. Αλλά η χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα φτάσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την εφαρμογή του νέου αυτού θεματολογίου. Τα χρήματα δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Η πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική όπως είπε ο προηγουμένως στο πρώτο πάνελ που είχαμε σήμερα. Οι πολιτικές είναι σημαντικές για να μπορέσουμε να κάνουμε την πιο καλή χρήση των πόρων για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους και να τους χρησιμοποιήσουμε εκεί που χρειάζεται και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική τους χρήση. Από αυτά που ακούσαμε σήμερα λοιπόν θέλω να υπογραμμίσω μία μονάχα σημαντική πτυχή που αναφέρθηκε η Αμίνα Μωαμέτ τόνισε την ανάγκη να έχουμε αξιόπιστους στατιστικούς δείκτες και μηχανισμούς εποπτείας και παρακολούθησης για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε την πρόοδο και να δούμε που χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Όλα αυτά θα είναι κέρια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και μεταξύ χωρών και μέσα στις χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα είναι πολύ σημαντικά γιατί αυτός γίνεται πια και ένας νέος στόχος καταπολέμησης της ανισότητας, στόχος 10. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί αν δεν έχουμε αξιόπιστους στατιστικούς δείκτες, το ευαλωτότερο τμήμα της κοινωνίας θα είναι αόρατο και θα είναι απόκληρο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι κανένα δεν θα μείνει έξω από την ανάπτυξη και να εστιάσουμε σε πιο αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός για την παρακολούθηση στο επίπεδο αυτό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σάιμον Μάξουελ, ο οποίος είναι ερευνητής του Ιδρύματος για την ε, Ανάπτυξη στον Τρίτο Κόσμο και πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Δεξαμενών Σκέψεων ο κύριος Μάξουελ έχει δουλέψει για την για την Εθνό και έχει εργαστεί και στη Βολιβία και στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ. Μετά θα δώσω το λόγο στον πρεσβή κύριο Πάτρικ Γκόμις, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της ομάδος ΑΚΕΠ. Ο κύριος Γκόμις έχει εργαστεί εδώ και 35 χρόνια με τις διάφορες αυτές, με τους φορείς των χωρών ΑΚΕ και έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών ήταν ε, επίσης σύμβουλος για το Ίδρυμα Τροφιμικής Ασφάλειας της Καρικόμ και είναι και στο κέντρο διαχείρισης και Δίκτυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάξουελ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά περίπου. Ευχαριστώ Ελή σκεφτόμουν τις επιπτώσεις αυτής της συζητήσης για εσάς τους Ευρωβουλευτές ή που δουλεύετε για το Ευρωκοινοβούλιο και για μας που είμαστε οι θειασότες σας στον κόσμο. Υπάρχουν τέσσερα συμπεράσματα που βγάζω εγώ από τη συζήτηση και στις επιπτώσεις τη ε, της συζήτησης αυτής θα επανέλθω μετά. Προφανώς εδώ πρόκειται για ευκαιρία εορτασμού. Ε, έχουμε αυτές τις δύο επιτροπές, ΔΕΒ και Περιβάλλοντος, που συνεργάζονται. Επίσης, είναι θαυμάσιο το ότι έχουμε ένα πλαίσιο, ένα checklist, όπως είπε η Αμήνα, που κάνει τα εξή δύο πράγματα. Συνδέει την ανάπτυξη και το περιβάλλον και το βορρά με τον νότο. Αν ήσασταν Πρωθυπουργό και έπρεπε να υπογράψετε αυτό το έγγραφο και σα έλεγαν ότι θα φυλακιστείτε αν οι στόχοι αυτοί δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρι το 2030 και ακόμα και μετά την, την πάση της Πρωθυπουργία σας θα σας βάζαν ε, στη φυλακή εάν δεν υπογράφατε, Δεν τους υπογράφατε γιατί είναι, παρά είναι φιλόδοξοι, παρά είναι ευρύς και περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούν με τίποτα να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Οι θάλασσε είναι πεντακάθαρες. Μέχρι το 2030 θα εξα, εξαλειφθούν όλα τα, όλες τις προβληματικές ουσίες, μέσα 15 χρόνια δηλαδή. Καλά, είναι ευκαιρία εορτασμού, αλλά σήμαστε είμαστε και λιγάκι ρεαλιστές για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Και αυτή η στόχη είναι απλώς ένα benchmark, είναι ένα ιδεατό. Γιατί όπως είπε και η Αμίνα, ε, κάθε περιοχή, κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει τη δική της προσπάθεια με αυτούς τους στόχους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη στιγμή που αυτοί οι στόχοι υπογραφούν, η αστυνομία των στόχων αυτών θα σας χτυπήσει την πόρτα γιατί δεν θα είσαστε νομοταγείς. Θα, μας, θα σας πει, α, είναι τα μέσα του 2000 ας πούμε 19 και εσείς δεν έχετε καθαρίσει τις θαλασσές σας. Επομένως πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι λέμε στο κοινό. Είναι φιλόδοξα αυτά τα πράγματα, είναι πλήρη, είναι, μ, βάζουμε τον πέχη ψηλά. Ε, δεν θα πρέπει να τα παίρνουμε και κατά γράμμα, έτσι. Φιλοδοξία υπάρχει, αλλά να μην τα παίρνουμε και τη μετρητή. Το δεύτερο, που θα είναι ακόμα πιο αμφίσιμο, αυτό που έχει σημασία το 2015 σήμερα δεν είναι η Αντισαμπέμπα, δεν είναι η Νέα Υόρκη. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι το Παρίσι. Γιατί εάν δεν έχουμε μια καλή κλιματική συμφωνία στο Παρίσι, τότε δεν έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, γιατί δεν θα έχουμε καμία περίπτωση να τους υλοποιήσουμε τους στόχους. Τι, τι σημαίνει λοιπόν τώρα καλή συμφωνία στο Παρίσι για το κλίμα. Κάποιοι θα έχετε ε, διαβάσει τον οδηγό ας πούμε για όσους κάνουν πεζοπορίες. Ε, ένα, μια, υπάρχει μια νουβέλα ας πούμε με κομικού περιεχομένου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο προπολογισμό που έχουμε για τα αέρια του θερμοκηπίου το 2013 είναι, ή μάλλον έχουμε 42 ε, γιγατόνους όριο. Είναι ε, ο όγκος της Μαύρης Θάλασσας, έτσι. Εάν λάβετε υπόψη όλες τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει, πολλές από τις οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί, τότε η εκτίμηση για τα αέρια των θερμοκηπίου το 2030 είναι 57. Εάν στο Παρίσι λοιπόν δεν δεσμευτούμε να υλοποιήσουμε τους, τους 42 γιγατόνους ε, μέχρι το 2030, δεν θα υπάρξουν βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι. Θα πρέπει να εστιάσουμε την πολιτική μας δράση και την εκστρατεία μας, όχι μόνο στο πλαίσιο των στόχων, που είναι η τελική, ας πούμε, η κατακλίδα, αλλά ε, σε συγκεκριμένα επιτεύγματα στο Παρίσι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Τώρα, αυτό συνδέεται με το τρίτο σημείο που θέλω να πω οι πολιτικοί και όσοι υποστηρίζουν θα πρέπει να σκεφτούν λιγάκι τη χορογραφία όλων αυτών των ε, διασκέψεων. Πώς συνδέονται και πώς θα φτάσουμε στη συμφωνία. Και στην Αντισαμπέμπα φυσικά και στη Νέα Υόρκη, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στο Παρίσι. Οι διαπραγματευτές ε, θα πρέπει να ξέρουν ποιοι είναι οι μοχλοί που θα χρησιμοποιήσουν. Ο βασικός μοχλός αλλαγής για να υπάρξει μια παγκόσμια συμφωνία δεν θα είναι οι αντιπολεπτομέρειε τη διατύπωση και αν θα υπάρχει ας πούμε στα αναπαραγωγικά δικαιώματα, η αναφορά στα αναπαραγωγικά δικαιώματα ή η δίνα αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά υπό αυτή την έννοια ο Σαρτ είπε το πιο σημαντικό πράγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε γραπτό να φτάσει το 0,7% για το, μέχρι το 2030 και το 0,33 για τα νέα ε, κράτη-μέλη. 50 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Κάτω από αυτό που είχαμε υποσχεθεί στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ, εν αυτή την περίπτωση, θα να τις συζητήσεις. Αν ήμουν ε, αναπτυγμένη χώρα, δεν θα έκανα μεγάλες υποσχέσει, θα είναι μεγάλε υποσχέσει στην αμπέμπα, θα τι κρατούσα για αργότερα. Νέα Υόρκη, Παρίσι κτλ. Τέτοιο, τέταρτο σημείο. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων για το κλίμα είναι ότι οι χώρες θα πρέπει να δώσουν τις ε, εθνικές συνεισφορές τους, που είναι οι δεσμεύσεις για τους στόχους ε, του 42 γιγατόνων μέχρι το 2030. Κάθε χώρα θα πρέπει να έχει τέτοιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δικές της με αρκετά ψηλούς και φιλόδοξους στόχους για μια κλιματική δράση μέχρι το 2030. Γιατί δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για τους ε, αναπτυξιακούς στόχους. Αντί να έχουμε αυτό το τόσο φιλόδοξο πια πλαίσιο, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο όμως να εφαρμόσουμε, αλλά σε κάποιες χώρες δεν θα είναι δυνατόν, σε κάποιες ναι, αλλά σε κάποιες χώρες γιατί να μην έχουμε εθνικές συνεισφορές στους βιώσιμους αντιψηφιακούς στόχους και ας έχουμε ε, εθνικές ας πούμε ε, μελέτες για να δούμε αναχώρα μπορούμε να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα κτλ. Μπορούμε να αυξήσουμε κάθε χρόνο σε σχέση με τον ε, να πούμε τόσο τα εκατό του ΑΕΠ μας για αυτή την προσπάθεια. θα πρέπει αυτός, αυτή η ατζέντα να γίνει πραγματική, ειδικά όσοι δίνουμε αυτή τη μάχη στο μέτωπο. Αυτοί είναι οι τέσσερις ε, στόχοι, ας ε, τους ε, καλωσορίσουμε, αλλά ας αναγνωρίσουμε και τους περιορισμούς, ας αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος εξάλληψης της ανθρωπότητας, ας δούμε τη χορογραφία εδώ το 2015 που έχει σημασία και τι θα κάνουμε μετά ως Ευρωπαίοι. Υπάρχουν τρία-τέσσερα πραγματάκια, τρία-τέσσερα διδάγματα που μπορούμε να μάθουμε. Καταρχά, το θέμα τη χορογραφία, ε, τη ενορχήστρωση είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε λεφτά, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε και άλλα μέσα εφαρμογή που υπάρχουν στην ατζέντα τη Αντισαμπέτα. Τεχνολογία. Ο κύριος Κίνγκ, ο βασικό ε, ε, για αυτά τα θέματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτείνει κάποια πράγματα. Ε, αντίστοιχα ε, με το project Apollo για τις ανανεώσιμες όμως πηγές ενέργειας αυτή τη φορά. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να προσφέρουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, και κάτι άλλο. Κάθε μη κυβερνητική οργάνωση στις Βρυξέλλες ε, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει βγει στους δρόμους ε, για να ζητήσει από τη χώρα της να υλοποιήσει τι τις δεσμεύσεις αναπτυξιακής βοήθειας. Ας σκεφτούμε λοιπόν την ενορχήστρωση ας σκεφτούμε την προσφορά που θέλουμε να κάνουμε και ας α, πετύχουμε αυτές τις συμφωνίες τώρα, το 2015. Επίσης, κατ' επανάληψη έχει τονιστεί ότι είναι μια ατζέντα που είναι εσωτερική και διεθνής. Εθνική για μας, αλλά αφορά και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι το σχέδιο δράσης. Νόμιζα ότι ήταν ενδιαφέρον που η Κομισιόν μίλησε για το κόστος ε, των ε, επιδοτήσεων στις, στα ορυκτά καύσιμα, καύσιμα στις αντισώμενες χώρες. Το είπε. Αλλά δεν είπε τίποτα για το κόστος ε, των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα που δίνουμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησε μόνο για τι ανεπιστώμενε χώρε. Ε, ξοδεύουμε 88 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδο... επιδοτήσεις ε, και διερεύνηση ας πούμε ορυκτών πόρων που ίσως δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε. Ε, που δεν θα έπρεπε να εκμεταλλευόμαστε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε εσωτερικά για τους αναπτυσσόμενους ε, στόχους συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος. Μιλάμε πάρα πολύ για την Ευρώπη 2020. Υπάρχει μια διαδικασία αναθεώρηση ε, για το Ευρώπη 2020. Εμεί χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα Ευρώπη 2030. Γιατί μιλάμε για το πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων. Α έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα Ευρώπη 2030. Αυτέ οι δύο επιτροπές είναι στο κατάλληλο σημείο για να παίξουν ηγετικό ρόλο και να μας πούν τι είδου βήματα πρέπει να λάβει η Ευρώπη εσωτερικά και εξωτερικά σε, όλους, σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής αυτής της πολιτικής μέχρι το 2030. Ένα από τα διδάγματα που μάθαμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ είμαι ειδικό σύμβουλο στην Επιτροπή Ανάπτυξη που μιλάει για την αναπτυξιακή συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου η αναπτυξιακή συνεργασία αφορούσε το να φτιάξουμε κέντρα υγεία στην Τανζανία. Τώρα θέλουμε να δώσουμε δημόσια αγαθά α, διατομιακά. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε μια αναπτυξιακή επιτροπή και τα λέω ομά, έτσι, η οποία ασχολείται ε, με τον DCI, που δεν ασχολείται καθόλου με το EDF, γιατί το κάνει το Συμβούλιο Υπουργών και δεν ασχολείται με όλα αυτά τα εγκάθια θέματα, εμπόριο, φορολογία, ασφάλεια, μετανάστευση και φυσικά κλίμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται μια συζήτηση για το πώ το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δουλέψει διαφορετικά. Όχι μόνο με ειδικέ ακροάσει, αλλά με εξεταστικέ επιτροπέ, με συνεργασία. Ε, χρήσιμο θα ήταν ίσω να γίνει και εδώ αυτό. Και τέλο. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτή τη συζήτηση είναι ότι γίνεται λόγος ε, για στατιστικές, συγκρίσιμε. Τι πετύχαμε από τότε που είχαμε τους στόχου τη της χιλιετίας, τι αλλαγέ είχαμε στην υγεία κτλ. Αυτό που δεν κάνουμε όμως είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αλλάζει δραματικά λόγω της α, ανάπτυξης της Ανατολής, ε, της ανάπτυξης των τεχνολογιών, ο κόσμος το 2030 θα είναι τελείως διαφορετικό από το σημερινό κόσμο. Και αν ε, κάνουμε συζήτηση για τους αναπτυξιακούς στόχους και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τις δραματικές αλλαγές, ας πούμε, της ε, οικονομίας, δεν έχει νόημα. Εγώ δουλεύω 40 χρόνια ε, στον, τομέα της ανάπτυξης και βλέπω ε, ποια... Η Κίνα πόσο δραματικά αλλάζεται. Μιλάμε συνέχεια για την Κίνα, αλλά πόσα ξέρουμε για την Κίνα. Λίγα τελικά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τίγρη. Θα πρέπει ε, να μην αρκούμαστε απλώς σε, συγκρίσιμες, σε συγκριτικές μελέτες. Θα πρέπει να καταλάβουμε το γίγαντα αυτό, αν θέλουμε να μιλήσουμε για βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Ευχαριστώ σίγουρη ότι θα ακούσουμε σχόλια στη συνέχεια μετά από αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες σκέψεις. Ας περάσουμε... Εντάξει, περνάει η ώρα, αλλά έχουμε λίγα λεπτά. Θα δώσω το λόγο τώρα στο πρέσβη Κόμες για 10 λεπτά περίπου. Ευχαριστώ πολύ Μαργαρίτα. Θα αρχίσω λέγοντας ότι εκτός από τα ζήτω θα έπρεπε να ήμασταν και λίγο επικριτικοί όταν συζητάμε τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους θα πρέπει να το δούμε από πλευρά των 700 ε, εκατομμυρίων. Πώς έχει νόημα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να αρχίσουμε από αυτό που είπες και εσύ πριν, από τις ανισότητες. Και από πλευρά των χωρών και θα έλεγα ότι η παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα θα πρέπει να δεχτεί πρώτα απ' όλα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι δομές της ανισότητας είναι αυτές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ανισότητα δηλαδή οδηγεί σε έλλειψη συνοχής. Στα Ηνωμένα Έθνη, για παράδειγμα, έχουμε ένα προπολογισμό 10 εκατομμύρια. Ποιος το χειρίζεται. Υπάρχουν δαπάνες για πυρηνικά, για όπλα. Τι δίνει η ΕΚΟΣΟΚ των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι η Ευρώπη στο σύνολό της μπορεί να μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εξουσία και για τις ανισορροπίες που υπάρχουν όσον αφορά την εξουσία αυτή. Δημιουργούνται όπλα μαζικής καταστροφής και όχι μόνο όπλα γιατί υπάρχει και κυβερνοχώρος. Η Ευρώπη λοιπόν μπορεί να παίξει ρόλο στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες αυτές που υπάρχουν στον κόσμο ολόκληρο. Ένα δεύτερο θέμα που μας ε, απασχολεί είναι το πού βρισκόμαστε και το τι γίνεται με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες έχουν πετύχει το στόχο του 0,7, κάποιες άλλες όχι. Και όχι μόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και μη ευρωπαϊκών χωρών που θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν επίση να πετύχουν το 0,7%. Άρα λοιπόν στην Αδίσε πρέπει να δεσμευτούν και άλλες χώρες. Είναι μια υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί. Βέβαια θα περίμενε κανείς ότι στην Ευρώπη ο στόχος αυτός του 0,7% για την αναπτυξιακή βοήθεια θα έπρεπε να μπορεί να παρακάμψει τη γραφειοκρατία, τους μηχανισμούς αυτούς που δημιουργούν εμπόδια. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να διευκολύνουν το 0,7%. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ορίζονται άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν ως καθήκον την αναπτυξιακή αυτή βοήθεια. Αν όμως δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη με το σωστό τρόπο και δεν αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητά της, τότε είναι πιο δύσκολο να το πετύχουμε. Γι' αυτό και μίλησα πριν για τη συνοχή. Άμα θέλουμε συνοχή, πρέπει τη συνοχή να τη βάζουμε στην πράξη. Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι οι διπλωμάτες και άλλοι που συμμετέχουν σε διάφορες αποστολές πρέπει να έχουν ευαισθητοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η αναπτυξιακή βοήθεια συνηθίζουμε να μιλάμε για πολιτική βούληση και να λέμε ότι αυτή λείπει και γι' αυτό δεν πετυχαίνουν οι πολιτικές μας. Η πολιτική βούληση όμως από μόνη της αποτελεί μια λειτουργία. Αν δεν έχουν γίνει αρκετά από την κοινωνία των πολιτών, αν δεν έχουν γίνει αρκετά από αυτό που έλεγε ο Σάιμον, δηλαδή να κατεβούμε στους δρόμους και να ζητάμε, αν δεν υπάρχει κινητοποίηση, όχι μόνο μεταξύ πολιτικών αλλά στην κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα κλπ, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της ανάπτυξης. Και άρα έτσι δεν φτάνουμε στο 0,7%. Χρειάζεται συνδυτοποίηση δηλαδή. Η Επιτροπή αυτή, η Ανάπτυξης και η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουν, πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το εμπόριο. Και γιατί? Γιατί το εμπόριο και το κέρδος από το εμπόριο μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη του εμπόριου. Οι επενδύσεις επίσης είναι κάτι αναγκαίο. Θέλουμε λοιπόν επενδύσεις οι οποίες να στοχεύουν τους ε, φυσικούς πόρους με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με τέτοια νομοθεσία που να έχει σαν στόχο την πρόσθετη αξία. Ξέρετε ότι υπάρχει παράνομο χρήμα και αν το παρακολουθήσετε θα δείτε πού βρίσκονται οι εξορυκτικές βιομηχανίες, οι μεγάλες πολυεθνικές που ασχολούνται με τα ορυκτά, με τα δάση. Πρέπει να λογοδοτούν, πρέπει να έρθουν και να παρουσιάσουν το έργο τους και στο, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Ανάπτυξης για να δείξουν κατά πόσο όντω φροντίζουν για αυτή την προστιθέμενη αξία. Γιατί αλλιώς κορυνεύουν. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πολλά μπορούν να γίνουν για περισσότερη συνοχή στην πολιτική μας. Στη Γεωργία για παράδειγμα, αυτό το οποίο ζητάμε ως μηχανισμό για την σήμαση των προϊόντων, ζάχαρη για παράδειγμα, είναι πολύ αυστηρά. Αλλά τι γίνεται με το εμπόριο. Δεν έχει νόημα να δίνουμε αναπτυξική βοήθεια. Από την άλλη μεριά όμως οι εμπορικοί κανόνες να είναι απαγορευτικοί για τις αναπτυσσόμενες χώρες ή αν παραβιάζονται συνέχεια οι κανόνες για τους δασμούς. Μιλάμε για πρόσβαση, αλλά η πρόσβαση αυτή είναι θεωρητική τελικά. Η πρόσβαση πρέπει να είναι πραγματική. Γι' αυτό και γίνονται πολλές συζητήσεις γιατί το θέμα της προσφοράς δεν έχει αντιμετωπιστεί ούτε το θέμα της πρόσβασης. Και έτσι φτάνουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, στην τεχνολογία και στη χρήση της τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνολογίας. Πρέπει με τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους να καθίσουμε να ξανασκεφτούμε την αναπτυξιακή ατζέντα και να τη δούμε πολύ περισσότερο από την πλευρά των συμμετοχών των κυβερνήσεων για παράδειγμα, να δούμε την ιδιαιτερότητα των κυβερνήσεων, την πολιτική τους. Και έτσι και πάλι φτάνουμε σε αυτό το κύκλο όπου η ιδιαιτερότητα σημαίνει να καταλάβουμε ποιοι είναι οι εθνικοί μας στόχοι και πώς μπορούν να συμπληρωθούν και να ξέρουμε ότι οι δύο αναπτυξιακοί στόχοι μπορούν να βοηθήσουν. Θα σταματήσω εδώ παρόλο που θα ήθελα να μιλήσω για τα διάφορα επίπεδα και πώς έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Thank you, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόμις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση καταρχήν για τους βουλευτές. Μαρία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, να βάλετε τα ακουστικά σας πρώτα. Κύριε Γκάμις, κύριε Ευχαριστώ. έχω κάπως κριτική στάση απέναντι σε αυτά που είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι, τονίσατε να είναι κάπως εφαρμόσιμα τα πράγματα. Εγώ βλέπω πάντα να υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι, αλλά στην πράξη πάντα τα πράγματα είναι πολύ κάτω από τις προσδοκίες. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπατε. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερες πληροφορίες ώστε ω κοινοβουλευτικό να μπορέσω και εγώ να επιχειρηματολογήσω προς την κατεύθυνσή σα. Και κύριε Μάξουελ. Είπατε ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το 2020 αλλά και το 2030. Και γι' αυτό μου δημιουργήσατε το ερώτημα αυτό. Πώς εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις, τις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πώ θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τι στρατηγικέ που έχει ήδη αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030 στα πλαίσια των, ε, των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη. Πώ θα συνδεθούν τα δύο αυτά. Είναι έτοιμη η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να προσαρμόσουν του στόχου αυτού τη ανάπτυξη τη ε, Γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε πάντα ότι τα πράγματα προχωρούν παράλληλα. Έχουμε καλές ιδέες, έχουμε καλές προσπάθειες, οι οποίες όμως κινούν παράλληλα, κινούνται παράλληλα μεταξύ τους χωρίς να υπάρχουν σημεία σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Σλάιν. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας και θέλω να θέσω δύο ερωτήματα στον κύριο Μάξουελ, τον οποίο θέλω να συγχαρώ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρέμβασή του εγώ είδα να υπογραμμίζεται ότι εφέτος, που είναι ένα έτος τόσο σημαντικών αποφάσεων, η προσπάθεια επίτευξη συμβιβασμών είπατε ότι εμποδίζεται από το θέμα της χρηματοδότησης και από τα μέσα εφαρμογής των στόχων διώσιμης ανάπτυξης. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παρακολουθήσει τα θέματα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και εγώ είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω εδώ μια έκθεση της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζεται μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι πολύ πιο φιλόδοξη από αυτή που φαίνεται να διαγράφεται αυτή τη στιγμή με τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών. Το ερώτημα που ήθελα να θέσω τώρα είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα, εσείς είπατε ότι η διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα ενδεχομένως θα εξαρτιόταν η εφαρμογή των συμπερασμάτων της από τις ε, συνεδριάσεις της Νέας Υόρκης και του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι ή τουλάχιστον όχι ιδιαίτερα αισιόδοξοι όταν οι προοπτικές για την συνδιάσκεψη της Αντίσα Μπεμπα, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να δώσουν πραγματικούς καρπούς. Ποια είναι η προοπτική που υπάρχει για τη μελλοντική χρηματοδότηση. Το θέμα τώρα της προσθετικότητας, όταν μιλάμε για χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση του αγώνα για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει καταρχήν η αρχή που θα διέπει αυτές τις ενέργειες να είναι η προσθετικότητα. Υπάρχουν όμως κάποιοι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάπως τεχνητή αυτή η διάκριση μεταξύ της ανάπτυξης αφενός και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αφετέρου. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι αν έχει πράγματι νόημα να τονίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει πάντα προσεντικότητα και επομένως οι χρηματικές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της ένδυας αν θα πρέπει να εμποδιστούν από τους αντίστοιχους στόχους που μπορεί να έχουν ήδη αποφασιστεί σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ Πέδρο. Κύριος ε, Σιν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές για τις τόσο ενδιαφέρουσες απόψεις και σχόλια που μας έκανε. Για τον κύριο Μάξουελ. αναφερθήκατε στο ταξίδι σας στην Κίνα και το ρόλο που παίζει η Κίνα στα θέματα αυτά. Βλέπουμε σημαντική οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα η οποία τώρα μετριάζεται κάπως. Φαίνεται ότι η κινέζικη κυβέρνηση αρχίζει να επανεξετάζει το μοντέλο ανάπτυξή τη και κινείται περισσότερο προ την κατεύθυνση θεσμική αλλαγή. Και εδώ έρχομαι στο ερώτημά μου. Ένα από τα προβλήματα για του βιώσιμου στόχου ανάπτυξη που δεν έχει αντιμετωπιστεί από το πάνελ είναι ο στόχο που έχει να κάνει με την ποιότητα των θεσμών. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε εδώ λιγάκι. Γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι δεν είναι τόσο σημαντική η αναπτυξική βοήθεια. Αλλά το ερώτημά μου είναι, χωρίς περιεκτικά θεσμικά όργανα, χωρίς αποτελεσματικά θεσμικά όργανα, που είναι σημαντικά για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, η οποία διαφθορά κοστίζει στις αναπτυσσόμενες χώρες δέκα φορές περισσότερο από την συνολική και βοήθεια. Αν δεν αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κέρια θέματα τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν και στην Αντισαβέβα και στην Νέα Υόρκη και φυσικά έχουν να κάνουν και με την ΚΟΠ στο Παρίσι. θέλω να ξέρω λοιπόν αν μπορείτε να κάνετε κάποια σχόλια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο. Voorzitter, dank u Ευχαριστώ πρόεδρε. πρόεδρε. Δύο πολύ σημαντικοί ομιλητές αυτοί οι δύο τελευταίοι. Συμφωνώ και εγώ με την ερώτηση που τέθηκε στην αρχή, αλλά θέλω περισσότερες πληροφορίες από τη δικιά σας την πλευρά. Είπατε ότι τα χρήματα πρέπει να έρθουν από εκεί που, έπρεπε να, που πρέπει να έρθουν. Ναι, αλλά και θέλω να μου πείτε περισσότερα πράγματα και για τη σήμανση των προϊόντων. Τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες συγκεκριμένα για σας. Οπότε τάξη, διπλωμάτες, business class, αλλά εγώ θέλω πιο συγκεκριμένα να μου πείτε αυτό για τι είμαστε των προϊόντων. Και στον κύριο Μάξουελ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Λέτε ότι στην Ευρώπη πρέπει να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Έτσι είπατε. ότι κάποιες χώρες τηρούν τις υποχρεώσεις τους και κάποιες άλλες όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι στρεβλώνται και ο ανταγωνισμό μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και στη Γεωργία, στη χώρα μου. Όταν οι γειτονικέ χώρες δεν τηρούν ε, τις υποχρεώσεις τους για το άσωτο για παράδειγμα, για τα νητρικά. Αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε πώς μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα στη συζήτηση αυτή. Μπορούμε να συζητήσουμε για το κόστος. Βαλτικές χώρες και η υπόλοιπη Ευρώπη. Thank you. Thank you very much again. I would just... Ευχαριστώ. Πολύ σύντομη ερώτηση. Αναφέρθηκε το θέμα των ε, πρέσβη Γκόμες. Στην Επιτροπή ΤΕΔΗ δουλεύουμε πολύ τελευταίως για το θέμα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αναφέρατε το τεράστιο πρόβλημα των παράνομων χρηματοδοτήσεων. Οι παράνομες χρηματικές ροές ε, που φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι δεκαπλάσεις από την αντιξιακή βοήθεια. Αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό, κινδυνεύουμε αυτό που πει η δεξιά να το ακυρώνει η αριστερά. More specific if you can and to go a little more deep, deeper. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε λίγα περισσότερα από αυτού του θέματος. If I can begin with the earlier question. Να ξεκινήσω με το ερώτημα που θέσαμε οι συνάδελφοι. Και να δώσω περισσότερα στοιχεία. Τι προσανατολισμό έχουν οι άνθρωποι που αποστέλουμε σε αναπτυσσόμενες χώρες. Για αν καταλαβαίνουν το ρόλο της ανάπτυξης, αν ξέρουν από αυτά. Και είναι σημαντικό η λογοδοσία που υπάρχει ε, για τα θέματα της αναπτυξιακής βοήθειας. Τα κοινοβούλια ε, εγκρίνουν. Οι χώρες κάνουν αποστολές για να δουν τι γίνεται με αυτή τη βοήθεια. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο στέλνει, ας πούμε, ε, αντιπροσωπείες ε, για να παρατηρήσουν τις εκλογές. Αλλά η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και Εμπορίου ε, καλό θα ήταν να παρακολουθεί το πώς χρησιμοποιείται η αναπτυξιακή βοήθεια. Συχνά μιλάμε για την, το δυναμικό απορρόφησης. Το θέμα είναι τι δυνατότητα έχουν ε, οι φορείς ε, στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης όμως κτλ. λοιπά τι ικανότητα έχουν ε, να κινητοποιηθούν, κατά πόσο καθυστερούν, εάν έχουν την αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι εάν δεν κατανοούν, ας πούμε, τους εθνικούς α, αναπτυξιακούς στόχους. Στη δική μου χώρα, τη Γουιάννα, Υπάρχει μια εθνική στρατηγική, αλλά δεν ξέρω αν ο κόσμο καταλαβαίνει τη δομή τη στρατηγική αυτή, τι προτεραιότητε, το ρόλο τη αναπτυξιακή βοήθεια και το συντονισμό τη βοήθεια των δωρητών μεταξύ του UNDP κτλ. Ε, το Υπουργείο Γεωργία τη Δευτέρα, ο, ο βασικό, ο γενικό γραμματέα, α πούμε, ε, συναντάται ε, με διάφορου δωρητέ. Αυτό κατά πόσο συνδέεται με το τι κάνουν ας πούμε οι γεωργοί, ξέρω εγώ, ε, για να δούμε, να δούμε τι συμβαίνει. Να πάω τώρα στις παράνομες οικονομικές ροές. Το θέμα είναι πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Εάν υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, φυσικά θα πρέπει να δούμε το σύστημα δημόσιας διαχείρισης των οικονομικών. Ε, και το επιβλέπουν σύστημα. Μήπως ε, επιστρέφουν στην Ευρώπη αυτά τα λεφτά. Εάν κάπου ας υπήρχε μία ανάσχεση, θα σταμάτησε αυτό το φαινόμενο. Να δούμε επίσης και τα εμβάσματα που αποστέλλονται από νόμιμη εργασία και των μεταναστών που πάνε στι αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί υπάρχουν τρομερές επιβαρύνσεις. Τι θα κάνουμε επίσης με τις άλλες υπηρεσίες και φορείς όπου θα μπορούσαν, ε, τα λεφτά που στέλνουν οι μετανάστες, εάν ε, είχαν λιγότερες επιβαρύνσεις ας πούμε, να φτάνουν στον τελικό τους αποδέχτη και αν υπήρχε και ένας ελεκτικός μηχανισμός με τους κατάλληλους φορείς για να το ελέγχουν αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ κύριος Μάξουελ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω και εγώ σε μερικά από αυτά σημεία. Χαίρομαι με αυτό που είπατε για η ιδέα του να έχετε την αστυνομία των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης και το να υπάρχουν και εκθέσεις για το τι γίνεται. Εγώ είχα γράψει μια, ένα άρθρο λέγοντας ότι αν ο υπουργός για το ταχυδρομείο θα ήθελα να έχω παγκόσμιους στόχους για να, μπορούν, να μπορώ να ξέρω πότε παραδίδονται οι επιστολές. Θα πρέπει να υπάρξει ένα παγκόσμιο ε, στόχο για τη χρήση νητρικών αλάτων στα αγροκτήματα και μετά θα πηγαίνει η αστυνομία και θα πιάνει του παραβάτε. Δεν θέλω τώρα να συζητήσω την κινέζικη πολιτική. Μια φορά έχω πάει εκεί, δεν ξέρω αρκετά την Κίνα. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον στην παραμονή μου στην Κίνα ήταν να του ακούσω να μιλάνε για την ε, νέα φυσιολογική κατάσταση χαμηλή ανάπτυξη. 7% για αυτού είναι φυσιολογική ανάπτυξη. Για την Ευρώπη είναι βέβαια θαύμα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 χρόνια η οικονομία τους διπλασιάζεται σε μέγεθος. Δεν είναι λοιπόν κάτι το τετριμένο. Αυτό που θέλω να τονίσω λοιπόν για την Κίνα είναι ότι εμπλέκεται στην παγκόσμια οικονομία. Ο Τόμας Φρίμαν έγραψε ένα βιβλίο που λέει «Η γη είναι επίπεδη» και λέει ότι όταν εγώ ήμουν παιδί, έλεγε ο Τόμας Φρίντμαν, ο πατέρα μου μου έλεγε «Φάε το φαγητό σου, γιατί ένα παιδί στην Κίνα πεινάει αυτή τη στιγμή». Και λέει τώρα στα παιδιά του τελειώστε τα μαθήματά σας γιατί κάποιο παιδί στην Κίνα θέλει τη δουλειά σας. Νομίζω ότι υποτιμούμε τον αντίκτυπο των μεγάλων παγκοσμίων αλλαγών που συνδέονται τώρα με την ανάπτυξη της Κίνας. Και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα του πώς η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει στον 21ο αιώνα. Η παγκοσμιοποίηση δεν θα έπρεπε να είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, αλλά πολλοί τη βλέπουν έτσι. Αλλά σίγουρα ισχύει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια μακροχρόνια στρατηγική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την πολυπλοκότητά τους και αυτό περιλαμβάνει και την απασχόληση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύω λοιπόν πράγματι θα πρέπει να προκύψει μια στρατηγική για το 2030 η οποία να προέρχεται και από το πλαίσιο των βιωσίμων στόχων. Ας το κάνουμε αυτό και ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας για μια τόσο πλούσια περιοχή του κόσμου είναι δυνατόν να το πετύχουμε αυτό. Τι τίμημα πρέπει να πληρώσουμε, Πώ πρέπει να χρονίσουμε τις δράσεις πρέπει να κάνουμε. Πρώτα η ανάπτυξη και μετά η διανομή ή πρώτα η διανομή και μετά η ανάπτυξη. Πρώτα η παιδεία και μετά η υγεία ή πρώτα η υγεία και μετά η παιδεία. Πώ θα συνδέεται όλα αυτά σε μια πρακτική στρατηγική για την Ευρώπη είναι μια μεγάλη <clears throat> πρόκληση λοιπόν για την Κομισιόν. Εν τέλει για την χρηματοδότηση και τα θέματα της προσθετικότητα. Εγώ θυμάμαι την εποχή που λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα φαίνεται σαν όνειρο, ένα νοσταλγικό όνειρο του παρελθόντος, όταν νομίζαμε ότι μπορούμε να έχουμε επίτευξη των στόχων για αναπτυξιακή βοήθεια και πρόσθετα κονδύλια για την ε, αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. Προφανώ αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή χρηματοδοτείται από την αναπτυξιακή βοήθεια που ήδη δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να έχει. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στην Αντισαμπέμπα και να έχουμε έναν τρόπο που να καλύπτει και τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή, αλλά κέρια είναι η χρηματοδότηση. Τι μπορώ να πω εδώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι στοχευμένη η χρηματοδότηση και σύμφωνα με τον κύριο για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε πού δαπανά η Ευρώπη την αναπτυξιακή βοήθειας υποστηρίζω του να υπάρχει βοήθεια προς την Τουρκία αλλά αν δείτε την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια η, ο μεγαλύτερος ε, αποδέκτης είναι η Τουρκία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υποστηρίζουμε την Τουρκία όπως πρέπει για να έχει γραμμές υψηλής ταχύτητος και βρίσκεται μέσα στον κατάλογο των χωρών αποδεκτριών που έχει συμφωνήσει όσα αν είχαμε εστιάσει όμως σωστά την ανάπτυξη. Εκεί βοήθεια όπως πρόσθεσε να κάνει ο Πίμπαλξ για το DCI και το EDF. Τότε νομίζω να πάνε στις πιο φτωχές χώρες, τότε αυτό θα ήταν πολύ αποτελεσματικό. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από την προσπάθειά μας για τα φορολογικά καθεστώτα για να εξαλείψουμε την τιμολογική μεταφορά κτλ. Τι θα κάνουμε λοιπόν στην Αντίσα Μπέβα. Εγώ θα ήθελα η Ευρώπη να πει ότι το 2016 θα πετύχουμε το στόχο του 0,7%. Θα βρούμε τα 55 δισεκατομμύρια που χρειάζεται για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να πετύχουν <clears throat> τον στόχο αυτό. Αλλά θα δώσουμε αυτά τα λεφτά μόνο αν οι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες δεσμευτούν για την κλιματική αλλαγή. Τότε μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία. Θα δεσμευτούμε, αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε κάτι για να μειώσετε τις εκπομπές σας διοξιδίου του άνθρακος και αυτή είναι σημαντική διαπραγματεύσεων να γίνει φέτο πώς να εξορροπηθούν αυτές οι δεσμεύσει και είναι μια πραγματικά σημαντική πρόκληση για τι διαπραγματεύσει. Αν ήμουν διαπραγματευτής δεν θα άνοιγα όλα τα χαρτιά μου. Θα κρατούσα κάποιους άσους στο μανίκι. Θα έλεγα ότι του έχω, αλλά θα του άνοιγα μονάχα αν υπάρξει συμφωνία στο Παρίσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο μας ομιλητές για τα τόσο ενδιαφέροντα που μας είπαν. Δεν θα ολοκληρώσουμε εδώ. Με ιδιαίτερα τιμή θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο, στον Παύλο Βαγιάν, για να κλείσει την ακρόση αυτή. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, τις σκέψεις σας και ο Πάβο. Όντως έχω ένα τρένο πολύ σύντομα, γι' αυτό θα... να ξέρετε ότι θα φύγω σε λίγο. Εγώ πρέπει να κάνω μια mission impossible. Γιατί, γιατί πρέπει να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα μετά τη σημερινή συζήτηση, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Ακούσαμε όλες τις παρουσιάσεις, τη συζήτηση τα συμπεράσματα του καθενός και ο καθένας υπογραμμίζει κάτι διαφορετικό ως σημαντικό. Οπότε εγώ τρεις προσωπικές παρατηρήσεις έχω να κάνω και ελπίζω να συμφωνώ με τα δικά σας προσωπικά συμπεράσματα. Πρώτον, πολλοί ομιλητές υπογράμμισαν ότι οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να είναι οικουμενικοί, πρέπει να υπάρχει οικουμενικότητα να αποτελούν ένα σύνολο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω υπόψη μου του 92 τη διάσκεψη στο Ρίο. Τότε ήμουν επικεφαλής της φιλανδικής αντιπροσωπείας ως υπουργό Εξωτερικών και τότε για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να τα βάλουμε όλα μαζί. Περιβάλλον, ανάπτυξη. Όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος και όλες τις πτυχές της ανάπτυξης. Ο στόχος μας ήταν να εφαρμόσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις χώρες και τις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες και τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Τι έγινε έκτοτε? Χωρίσαμε το περιβάλλον από την ανάπτυξη. Χωρίσαμε τον περιβαλλοντικό τομέα στο κλίμα, την ε, τις πολιτικές ε, αποψήλωσης των δασών κλπ. Και όσον αφορά την ανάπτυξη και εκεί έγινε κάποιος κατακαιρματισμός. Τώρα θα έπρεπε να βάλουμε μαζί την ανάπτυξη και το περιβάλλον πάλι και να τα δούμε συνολικά. Αυτό είναι το πρώτο μου συμπέρασμα και συμφωνώ με τους ομιλητές που το τόνισαν στην παρουσίασή τους. Δεύτερον, μιλήσαμε για τους πυλώνες. Όταν συζητήσαμε για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, είπαμε ότι έχουμε 17 στόχους και 200 μέτρα. Όταν έχετε τόσες πολλές προτεραιότητες, είναι σαν να μην έχετε καμία. Θα έπρεπε λοιπόν κάπως να τους συγκεντρώσουμε. Ανακατηγορία μείωση της φτώχειας, καταπολέμηση των ανισοτήτων και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας. Τώρα, στη συνθετική εκθεσία ο Γενικός Γραμματέας χρησιμοποίησε την ιδέα των πυλώνων που είναι πολύ κοντά στις δικές μας τις ιδέες και νομίζω ότι όταν ολοκληρωθούν οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι και όταν φτάσουμε στην εφαρμογή τους θα πρέπει να τους συγκεντρώσουμε κάπως, να τους ταξινομήσουμε ώστε να γίνουν έτσι πιο αποτελεσματικές οι πολιτικές μας. Τρίτο συμπέρασμα όσον αφορά την εφαρμογή. Όλες οι πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν. Οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλα περιφερειακά όργανα, ο ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικέ οργανώσει, όλοι πρέπει να εφαρμόσουμε. Ο καθένα μα ατομικά πρέπει να εφαρμόσει του στόχου. Αλλά θέλω εδώ να υπογραμμίσω το ρόλο του συστήματο των Ηνωμένων Εθνών στην παρακολούθηση και την εφαρμογή. Βλέπετε, συντάσω μια έκθεση ιδία πρωτοβουλία στην, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΟΗΕ πώς να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Επιτροπή αυτή θα γνωμοδοτήσει νομίζω, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, έτσι. Εν περιπτώσει διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές συμμετέχουν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Το σύστημα λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματικό προκειμένου να μπορέσουμε και να εφαρμόσουμε τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Έχω κάποιες ζωσπαστικές ιδέες στην έκθεσή μου, θα τους δείτε κάποια στιγμή. Συνεπώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εξαίρετη ακρόαση, τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και την τόσο καλή συζήτηση. Ευχαριστώ.